Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. It is my pleasure, privilege ε, είναι τιμή μου και χαρά μου που εγκαινιάζω και σας καλωσορίζω στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλεια και Άμυνα που θα κρατήσει μια μισή μέρα και έχει πολύ ενδιαφέρουσα ημερήσια διάταξη. Χωρί άλλη λοιπόν καθυστέρηση θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας και να προτείνω πρώτα απ' όλα φυσικά την έγκριση της ημερήσια διάταξη. Μια και δεν βλέπω παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Καταρχήν να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων της 24ης και 25ης Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Η διορία για την υποβολή επιφυλάξεων στάσεων ή παρατηρήσεων ισχύει μέχρι τα τέλη της συνεδρίασής μας. Οπότε αύριο μέχρι το μεσημέρι έχετε διορία να υποβάλλετε προτάσεις ή παρατηρήσεις για τα πρακτικά, αλλιώς θα θεωρηθούν συγκεκριμένα. Και περνάμε στο πρώτο ουσιαστικό θέμα της σας διάταξης που περιλαμβάνει παρουσίαση της συμμετοχής ε, της Χιλής σε αποστολές ε, της κοινή πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας και τη συμμετοχή, συμπερίληψη της Χιλής στην, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ασφάλειας και Άμυνας. Εν ώψη των διαπραγματεύσεων για την εξεχρονισμό και ανανέωση της Συμφωνίας Σύνδεσης. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον εξοχότατο Ραούλ Φερνάντες, που είναι πρέσβης της Χιλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίσατε κύριε Πρεσβευτά. Και έχουμε και έναν εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ. Είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μας στείλει κάποιον εκπρόσωπο από το Τμήμα Εταιρικών Σχέσεων και Συμφωνιών. Είναι ο κύριος Φρεντερίκ Μαντιουγό. Υπεύθυνο, όπω είπα, των εταιρικών σχέσεων και συμφωνιών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα έχουμε πρώτα απ' όλα την παρουσίαση της, εκ μέρους της Χιλής, μιας χώρας που συμμετέχει σε αποστολές ε, της ε, κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή τη Χιλή ε, είναι ουσιώδη σε τέτοιε επιχειρήσει και αποστολέ. Για παράδειγμα, συμμετέχει στην Αλθέα, στην επιχείρηση Αλθέα και μάλιστα μία αποστολή της υποεπιτροπής μας θα μεταβεί στο Σεράγεβο για να ε, εξετάσει αυτή την επιχείρηση, την Αλθέα, στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Η Χιλή για πολύ καιρό ήταν μία από τις πέντε εξωκοινωτικές χώρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση Αλθέα στη Βοσνία Ριζεγοβίνη και προηγουμένως στην ΑΕΤ και σε άλλες χώρες. Χωρίς άλλη θα δώσω το κόσμο, τον λόγο στον ε, πρέσβη της Χιλής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι μέλη της, Επιτροπής, ε, της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνα, ε, κύριε εκπρόσωπε της ΕΙΕΔ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, την κυρία Φωτίγκα, για την πολύ ευγενική πρόσκληση που μου έκανε να λάβω μέρο σε αυτή τη συνεδρίαση και μάλιστα σε τόσο σημαντική στιγμή για το μέλλον των σχέσεων Χιλή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χιλή είναι μια αξιοσέβαστη χώρα του Διεθνου δικαίου με έντονη πολυμερή προσέγγιση και πάνω από 60 χρόνια συμμετείχε σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσει. Η πατρίδα μου συμμετείχε ενεργά στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και σε διεθνή φόρα ε, για την ασφάλεια και την ε, ειρήνη. Συνέβαλε μάλιστα ενεργά στην διαφύλαξη της διεθνούς ε, ειρήνης και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την αμυντική πολιτική, έχουμε μια ευρεία πολιτική με βάση την αρχή της συνεργασίας στο πολυμερές σύστημα. Δεδομένου ότι τα εθνικά συμφέροντα της ασφάλειας και άμυνας συνδέονται αναπόσπαστα με την ειρήνη και την ασφάλεια του κόσμου. Γι' αυτό συμμετέχουμε ενεργά και είμαστε υπέρμαχοι της ε, διεθνούς ειρήνης. Θεωρούμε ότι οι ευθύνε μας ε, ως προς τη συνεργασία έχουν θεμελιώδη σημασία γιατί υπάρχουν κάποιοι παγκόσμιοι κίνδυνοι. Κανένα μέλος της διεθνούς κοινότητας ε, που είναι υπέρμαχος της ειρήνης, της ασφάλειας και του κοινού συμφέροντος δεν μπορεί να αποποιηθεί αυτή τη ευθύνη για συνεργασία. Η παγκόσμια συνεργασία είναι ένα κοινό καθήκον, συλλογικό, και αυτό και θα πρέπει και η δέσμευσή μας να είναι συλλογική. Η Χιλή είναι υπέρ των οικουμενικών αξιών και αρχών σε πολυμερείς φορείς συνεργασίας, προκειμένου να ενισχύσουμε τα διεθνή καθεστώτα ασφάλειας. Γι' αυτό από το 1949 τη στιγμή που συμμετείχαμε στην ειρηνευτική επιχείρηση στην Ινδία και το Πακιστάν, δώσαμε το παρόν σε πολλές χώρες, στην Καμπότζη, στην Ικαράγουα, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την ΑΕΤ μεταξύ άλλων. Και μάλιστα στην ΑΕΤ ήμασταν στη Μινούστα. Στείλαμε 10.000 προσωπικό σε 13 χρόνια. Και στη δεκαετία του 90 είχαμε ένα πραγματικό σημείο καμπής για τη Χιλή. Και από χώρα που στέλαμε μόνο παρατηρητές ειρηνευτικές αποστολές, περάσαμε στην ανάπτυξη και στρατιωτικών μονάδων σε επιχειρήσεις συνεργασίας με βάση τα κεφάλαια 6 και 7 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ε, γίναμε έτσι ένας ε, σημαντικός παράγος συνεργασίας ε, στη διεθνή ειρήνη. Η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας ε, ανάγεται στο 2004. Τότε η Χιλία αποφάσισε να λάβει μέρος στην επιχείρηση EUFOR Altea της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με πρωταρχικό στόχο την ε, επιτήρηση της εφαρμογής των ειρηνευτικών συμφωνιών του Dayton του 1995. Η παρουσία της Χιλής ε, στα Βαλκάνια ξεκίνησε το 2003 με τη συμμετοχή στις ΦΟΡ στην σταθερο... στα... σταθεροποιητική δύναμη του ΟΗΕ υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Η Αλτέα ε, συμμετέχει στην εκπαίδευση των ε, Βοσνίων και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της Βοσνίας Ριζεγοβίνης. Μάλιστα έχει λύνει η μόνη λατινοαμερικανική χώρα που μονίμως συμμετέχει σε μια ειρηνευτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα από την αρχή της ε, καθιστώντας μας ε, σημαντικό διεθνή φορέα υπέρμαχο της ε, ειρήνης. Και μάλιστα είχαμε μεγάλο αριθμό προσωπικού από τον Ιανουάριο του 2008 και μάλιστα προσθέσαμε και έναν επιπλέον αξιωματούχο στο εθνικό μας απόσπασμα εκεί. Και φάνηκε ο επαγγελματισμός και η ικανότητα των χιλιανών στρατιωτών και του χιλιανού προσωπικού που συμμετέχει στην επιχείρηση Αλτέα. Το 2014 ε, υπογράψαμε μία συμφωνία πλαίσιο διαχείρισης των κρίσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής ε, που τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2015 και αναφυσβήτητα αυτό αυτή η συμφωνία πλαίσιο είναι ένα επιπλέον βήμα πρόοδου στι διμερεί μα σχέσει με δημιουργία επαρκού νομικού πλαισίου που θα διευκολύνει τη συμμετοχή τη Χιλής και σε άλλε επιχειρήσει και ειρηνευτικέ αποστολές τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία τέτοιου χαρακτήρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει με Λατινοαμερικανική χώρα. Επίση, τον Απρίλιο του 2015, ευκαιρία του Συμβουλίου Σύνδεση. Ε, που έγινε στις Βρυξέλλες με προεδρία της κυρίας Μογκερίνη και με τον Εράλντο Μουνό τον τότε υπέξ της Χιλής. Ε, συζητήσαμε τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, κάτι που δείχνει πόσο σημαντική, σημαντικό γίνεται αυτό το θέμα στις διμερείς σχέσεις. Ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας Σύνδεσης Χιλής Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράψαμε το 2002, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Ε, ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2016 και φέτος το Φεβρουάριο ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος των σχετικών διαπραγματεύσεων. Και μάλιστα η επιτυχία της Συμφωνίας Σύνδεσης και για τη Χίλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διάφορους τομείς μας έφερε το 2013 να εκδηλώσουμε την ανάγκη και οι δύο πλευρές να εξυγχρονίσουμε τη συμφωνία. Είδαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι οι διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής εδράζονται στις ίδιες αξίες και αρχές και θα αποτελέσουν και τη ραχοκοκαλιά της νέας εξυγχρονισμένης συμφωνίας. Η σημασία του ανθρώπου, των οικομενικών αρχών και αξιών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας, της πάταξης των διακρίσεων, της ισότητας των δύο φύλων και της χειραφέτησης ε, ενδυνάμωσης των γυναικών, η διαφάνεια, η στήριξη της αηφόρου ανάπτυξης είναι βασικές αρχές που θα κατοχυρωθούν και στη νέα εξυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης. Θέλουμε να, δώσουμε, να προβάλλουμε περισσότερο την ε, αυτή συμφωνία και να θεσπίσουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα ε, διαμορφώσει τις μελλοντικές σχέσεις της Χιλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα οι τομείς που επιδέχονται μεγαλύτερη συνεργασία είναι ακριβώς ε, οι τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Και ναι, μεν στην παρούσα συμφωνία έχουμε κάποιες ακροθυγείς διατάξεις για, το θέμα, για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, κυρίως τα άρθρα 14 και 15 πραγματεύονται αυτά τα θέματα, θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα διεύρυνση τη συνεργασία στην ασφάλεια και στην άμυνα. Γι' αυτό και οι τρέχουσε διαπραγματεύσει θα συμπεριλάβουν μία σειρά διατάξεων για τον αφοπλισμό, μη εξάπλωση των όπλων, την διεθνή ασφάλεια, τον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση των μη παραδοσιακών απειλών όπως και της θερμοκρατίας, μικρά και ελαφρά όπλα και άλλα συμβατικά όπλα, διαχείριση των διεθνών κρίσεων και ούτω καθεξής. Βέβαια, ακόμα εκκρεμούν οι διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουν τα συμβαλώμενα μέρη να επιτύχουν ευρεία και εις βάθος συμφωνία σε όλες τις επιμέρους αυτές τις πτυχές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Excellency, thank you very much indeed. Now... Σας ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά. Θα ήθελα τώρα να δώσω στον το λόγο στον κύριο Μαντουρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε σχέση με την προηγούμενη ομιλία του πρεσβευτού Φερνάντες για τα γεγονότα που συζητάμε εδώ, δεν έχω πολλά να προσθέσω, απλά και μόνο να υπογραμμίσω τη σημασία και να τιμήσω τη σημασία της συμβολής της Χιλής που από το 2004 συμβάλλει συνεχώς στις επιχειρήσεις μας όπως αυτή στην Βοσνία την ολτέα. Από το 4 λοιπόν έχουμε 500 άτομα, πάνω από 500 άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν την αποστολή και φέτος είδαμε ότι το Δεκέμβρη είχαμε 15 ακόμα άτομα από τη Χιλή που συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή έχουμε μια συμφωνία συμμετοχής, συμφωνία πλαίσιο για την επιχείρηση αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόγραψε σήμερα 18 τέτοιες συμφωνίες. Η πρώτη υπογράφηκε και επικυρώθηκε στη συνέχεια με την Χίλη όπως είπαμε και έχουμε υπογράψει και μία παρόμοια συμφωνία με την Κολομβία αλλά δυστυχώς η συμφωνία αυτή δεν έχει ακόμα επικυρωθεί. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι αυτή η συμφωνία πλαίσιο συμμετοχή έχει μια πολιτική διάσταση αλλά και μια επιχειρησιακή διάσταση και επιτρέπει την συμμετοχή της χιλής στις επιχειρήσεις και αποστολές μας της ΚΠΑ. Βεβαίως στόχος μας είναι αυτή η συμμετοχή από το 14 ανισχύει τη συμμετοχή της Χιλής και σε άλλες αποστολές και επιχειρήσεις. Έχουμε επαφές για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή της Χιλής σε αποστολές και επιχειρήσεις όπως την ε, Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Έχουμε λοιπόν όλες ε, αυτές οι επαφές και για την επιχείρηση Αταλάντα. Είναι διερευνητικές επαφές, αλλά δυστυχώς επειδή έχουμε περιορισμούς οικονομίας δεν μπορέσαμε να επιτρέψουμε πλήρη συμμετοχή της χιλής και άλλες ε, επιχειρήσεις της ε, Αυτά. Για το μέλλον είναι σημαντικό να καθορίσουμε το μέλλον των σχέσεών μας με τη Χιλή στα πλαίσια της ε, μεταρρύθμισης των πολιτικών μας όσον αφορά το πλαίσιο εταιρικών σχέσεων για θέματα ασφάλειας και άμυνας όπως είπε και η Υπατη εκπρόσωπος Έχουμε και τη συζήτηση λοιπόν για, αυτό, για, για τη μεταρρύθμιση αυτού του πλαισίου συνεργασία. Βεβαίω εμεί θα συνεχίσουμε τις προσπαθίε μας προ αυτή την κατεύθυνση. Δύο εργασία για το μέλλον. Διερευνητικέ επαφέ και διάλογο όσον αφορά τα θέματα άμυνα και ασφάλειας. Το δόγμα που επιδιώκουμε μέχρι σήμερα ήταν το συστηματικά κάθε φορά που έχουμε μια επιχειρησιακή συνεργασία, να καθορίσουμε ένα διάλογο όσον αφορά τα θέματα αυτά ασφάλειας και άμυνας με τρίτες χώρες που έχουν συνάψει με εμά ε, συμφωνίες πλαίσιο και μια δυνατότητα για το μέλλον θα ήταν το να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών κάτι το οποίο βεβαίω θα ανοίξει ένα νέο χώρο συνεργασίας μεταξύ της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως θα θέλαμε να προβλέψουμε τη συμμετοχή ως παρατηρητών αυτών των εταίρων μας στις επιχειρήσεις μας και να ενισχύσουμε επίσης και τις δυνατότητες εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Χιλής. Όπως υπόθηκε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την αναθεώρηση στην οποία προχωρήσαμε σχετικά με τη νέα συμφωνία σύνδεσής μας και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων. Αναγνωρίζοντας βεβαίως το όλο και πιο σημαντικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και Χιλής στα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντουρού. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συμμετέχοντες. Ο κ. καλά θα ήθελε να συμμετάσχει νομίζω. Να συμβάλλει. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως θέλω. Θα μιλήσω γερμανικά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρέσβη, για την παρουσίασή σας και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, ακούγοντας κανείς την ομιλία σας, ε, κύριε Πρέσβη, πραγματικά κανείς δεν ε, αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται η Χιλή στο χάρτη. Δηλαδή θα είχε την αίσθηση ότι είτε είναι μέλος είτε είναι υποψήφιο προς προσχώρηση μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όπως είχα πει και κάποτε στο παρελθόν, ε, εάν δηλαδή βρισκόταν στα ανατολικά της Γρυλανδίας και όχι στα δυτικά της Γρυλανδίας ο Καναδάς, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η γεωγραφική απόσταση ωστόσο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής ε, γεφυρώνεται ε, χάρη ακριβώς στην, στη συγγένειά μας και σε ό,τι αφορά τις βασικές μας θεμελιώδεις αξίες. Και δεν το λέω αυτό απλά έτσι. Πραγματικά θεωρώ πως ισχύει και έχει αναπτυχθεί ένα σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα καθώς και μια σταθερή οικονομία ε, και κατά συνέπεια υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές ε, προϋπαθέσεις ε, καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών σε μια σειρά από τομείς. Και γι' αυτό σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες αυτής εδώ της Επιτροπής θα ήθελα και θα ήταν πολύ καλό να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας. Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχουν ενημερώσει, υπάρχει και ένα πλανητάριο εκεί, έτσι, ένα τηλεσκόπιο, νομίζω στη Χιλή, λόγω ακριβώς της καθαρής ατμόσφαιρας ε, τη Αντι, το οποίο έχει πάρα πολύ πάρα πολύ ψηλή ευκρίνεια. Ίσως ε, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αναπτύξουμε μια συνεργασία σε ό,τι αφορά το δορυφορικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εδώ εγώ δεν έχω να κάνω ερωτήματα δίνω ερεθίσματα για σκέψη ως προς τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη συνεργασία, εντατικότερη συνεργασία. Ε, είναι δηλαδή πολύ θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εταίρους οι οποίοι βρίσκονται μακριά της ε, γεωγραφικά, αλλά με τους οποίους ε, είναι δυνατόν να υπάρχει μια ακόμα καλύτερη συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρεσβευτή για την παρουσία του που μαρτυρεί κάτι που ήδη δυστυχώς γνωρίζουμε, ευτυχώς γνωρίζουμε. Δηλαδή αυτή η προσήλωση ξεπερνά τους ιδεολογικούς φραγμούς και η πρόεδρος Πινέρα που κλέφτηκε πρόσφατα έχει αυτή την αντίληψη σχέση με αυτά τα θέματα και τις σχέσεις με την Ένωση και θα ήθελα εκ μέρου του ΕΛΚ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον αδελφού Κάλερ να αναγνωρίσω την προσπάθεια αυτή και τη συμβολή της, Χι, σε διάφορες επιχειρήσεις ευρωπαϊκές. Έχουν λοιπόν θαυμάσια σχέσεις οι οποίες πηγαίνουν πέρα των σχέσεων που έχουμε με πολλές άλλες χώρες της Ένωσης. Να πω και στον κύριο Μαντουρό ότι τον ευχαριστώ για, τη, για τα λόγια του που μαρτυρούν την συνεργασία μας με τη Χιλή και να πω επίσης ότι εδώ πέρα έχουμε αυτά, αυτά τα ακτικόλεξα και τι να σας πω, καλή τύχη γιατί δείχνει ακριβώς το μέγεθος των επιχειρησιών μας, των δραστηριοτήτων μας. Έτσι. Θα πρέπει να ε, να σας πω ότι το κάνω αυτό, το λέω αυτό για να συμβάλλω ακριβώς στην σαφήνεια αυτού του ευρωπαϊκού λεξιλογίου, ιδιαίτερα προς τους ευρωπαίους πολίτες μας. Ε, σχόλιο επικοδομητικό αυτό. Αυτά, τίποτα άλλο και να ευχαριστήσω τον ε, Περσβευτή για τις προσπάθειες τις οποίες πραγματικά αναγνωρίζουμε όλοι. Και μας τη ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω τις δικές μου ερωτήσεις ως τακτικό μέλος. Το πρώτο ερώτημα αφορά και τους δύο διακεκριμένους ομιλητές μας και αφορά τις διατάξεις των μελλοντικών συμφωνιών σύνδεσης σε τομείς συνεργασίας όπως ιδιαίτερα τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση και αν γίνεται θα ήθελα να ακούσω κάτι παραπάνω σε σχέση με τις ενδεχόμενες διατάξεις για τις προσδοκίες για τη συνεργασία αυτή ενός εσχυλής για αυτά τα θέματα. Και δεύτερον, προς τον Προσβευτή Φερνάντες, να πω ότι βάσει της εμπειρίας της Χιλής στην Βοσνία Ζεγοβίνη πώς αποτιμάτε την τωρινή κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταστροφή όπλων και την στρατιωτική συμμετοχή. Έχετε το λόγο εσείς. Να απαντήσετε με την ίδια σειρά. Πρώτα ο κύριος Περευτής και μετά ο κύριος Μοντιγού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για τον κύριο Κάλερ να πω ότι ευχαριστώ για το σχολείο του, όπως και τον κύριο Λόπες Αστορίθ. Η Ευρώπη συμμετέχει στο αστρονομικό παρατηρητήριο και συνεργαζόμαστε στενά και έντονα με τις Ευρωπαϊκέ αρχές για αυτό το θέμα αιχμή. Και χαιρόμαστε πολύ που υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ της ε, Χιλής και της Ένωσης σε αυτό το ε, χώρο, σε αυτό το πεδίο. Για τη μη διάδοση των όπλων, θέμα σημαντικό των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του πολιτικού πλαισίου συνεργασία και σε σχέση βέβαια με τι απειλέ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μα και έχουμε μια κοινή οπτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να πιστεύω τώρα σε λεπτομέρειε σε σχέση με το τι σημαίνει ή τι σημασία έχει το τωρινό κείμενο, γιατί βρισκόμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσει. Αλλά είμαι βέβαιο ότι θα καταλήξουμε σε έναν καλό, ισχυρό και εξυγχρονισμένο κείμενο. Τώρα για τι επιπτώσει τη συμμετοχή μα στην Βοσνία Ερσεγοβίνη, να πω καταρχά ότι εκτός από τη συνεργασία που προποθέτει η δέσμευση της χιλής θα πρέπει να πούμε ότι η εμπειρία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τις στρατιωτικές μας δυνάμεις. Το γεγονό και μόνο ότι με στρατιωτικές δυνάμεις άλλων χωρών είχαμε συνεργασία και η εμπειρία, αυτό αποτελεί κάτι το πολύ σημαντικό από μόνο του. Χαιρόμαστε πολύ για αυτό που κάναμε στη Βοσνία Ερσεγοβίνη και θεωρούμε ότι λείπουν ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να συνεχίσουμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαντιγό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να επανέλθω στην ερώτηση του κυρίου Λόπες Ιστορής για τα ακρονίμια. Λυπάμαι που δεν ήμουν σαφής προηγουμένως. Ε, εγώ δεν είχα την αίσθηση ότι έκανα κατάχρηση των ακρονιμίων και των αρχικών στην ομιλία μου. Ε, για να με καταλαβαίνουν μόνο οι επαείοντες σε θέματα κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ή όσοι μετήχαν ε, στο συμφωνία πλαίσιο, αλλά είμαι στη διάθεση να εξηγήσω οποιασδήποτε απορίες. Όχι, δεν ε, αναφέρθηκα στην ομιλία σας, αλλά στον τίτλο σας. Είπα ότι ο τίτλος σας είναι πολύ περίπλοκος καμία σχέση με την παρουσίαση, ήταν ε, εξαιρετική. Απλώς βλέποντας ε, τον τίτλο, εντάξει το EAS το καταλαβαίνω, είναι η ΕΕΔ, e Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα υπόλοιπα αρχικά του τίτλου σας δεν κατάλαβα. Ναι, εμείς είμαστε επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των συμφωνιών εταιρική σχέσης ε, σε θέματα κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και ασχολούμαστε με την τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών πλαίσιο και στα πλαίσια της αναθεώρησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης το τμήμα μας έχει αναλάβει εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θεσπίσει αυτή τη νέα πολιτική εταιρικών σχέσεων και αυτό είναι το πλαίσιο που ρυθμίζει τις εργασίες μας. Αυτά ως προς τη θέση μου και το τις αρμοδιότητές μου και τις ευθύνες μου. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος που να ζητάει το λόγο. Οπότε θα ήθελα όλοι μας να χειροκροτήσουμε εδώ τους ομιλητές μας για την ε, πολύ περιεκτική τους παρουσίαση. Ευχαριστούμε τον αυτοξοχότητα τον ε, κύριο Πρέσβη. για την παρουσία του σήμερα εδώ, προκειμένου να μας κοινοποιήσει τις θέσεις του σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία μπορούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Should we wait? Well, we have 20 minutes. We can make a break of 20 minutes. Yeah. Because Mr. Yeah. Colleagues, uh, next point. Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο στις 10 η ώρα. Δηλαδή, ε, την ε, παρουσίαση της ε, έκθεσης ΠΑΕΤ σε ό,τι αφορά την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε τότε στις 10. Ναι, Πρόεδρε. Είχε προβλεφθεί να ξεκινήσει στις 10 αυτή η έκθεση. Γιατί παρευρίσκομαι, είμαι σκιώδη συζητητής από την πλευρά του ΕΛΚ. Οπότε, πρόεδρο, ναι, αλλά πρόκειται για την έκθεση του συναδελφού Πάιτ. Σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολλοί ομιλητέ στο πλαίσιο του προηγούμενου σημείου τη μερική διάταξη, γι' αυτό τελειώσαμε λίγο νωρίτερα. Colleagues, please be seated. Thank Καθίστε σας παρακαλώ συνάδελφοι και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Το επόμενο λοιπόν σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η εξέταση του σχεδίου έκθεσης ε, σε ό,τι αφορά την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Ο κ. Σούρμας Πάετ από τους φιλελεύθερους είναι ο μας για αυτήν την έκθεση και καθώς ε, παρευρίσκονται ε, και περισσότεροι από τους ασκιώδες εισηγητές ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε την εξέταση αυτού του σημαντικού ζητήματος, δηλαδή του σχεδίου έκθεσης για την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Ο λόγος στον κύριο Πάτ Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Όπως όλοι γνωρίζαμε, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των, ε, του διεθνούς ε, γίγνεσθε και η δική μας έκθεση εστιάζει στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κυβερνοχώρο. Ε, καθώς βέβαια ή μάλλον παρότι συνεχίζει να αποτελεί βασικά ε, εθνική αρμοδιότητα η άμυνα στον κυβερνοχώρο, καθώς ε, λόγω της φύσης ε, του εγκλήματο στον χώρο δεν ε, πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει το κάθε κράτο μέλο μόνο ε, Χρειάζεται μια συνεργασία και εδώ μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είδαμε στο πλαίσιο του σχεδιασμού τη Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική κατά τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν προσπάθειες και στο επίπεδο του χώρου. Για παράδειγμα, έχουμε τις τελευταίες ε, πρωτοβουλίε τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα για την υποστήριξη αντίστοιχων προσπαθειών. Δύο project έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία ε, αντίδραση, αλλά περισσότερα θα πρέπει να γίνουν. Θέλουμε δηλαδή να υπάρξει περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα επιτελεία του για το χώρο, για να επιτύχουμε περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών, περισσότερη εκπαίδευση αλλά και περισσότερη επιχειρησιακή υποστήριξη. Επίση, θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άνιμο για αυτόν τον σκοπό. Οι ε, αποστολέ ε, τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα βασίζονται σε αντίστοιχα ε, συστήματα πληροφορική τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικού στόχου για επιθέσει. Άρα λοιπόν κάποια τα οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε θα πρέπει να αποτελούν τμήμα τέτοιων ε, επιχειρήσεων ε, κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνα. Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αυξηθεί και αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη ε, στο πλαίσιο αυτών των αποστολών. Αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτό το τομέα είναι η έλλειψη εμπειρογνωμόνων, ειδικών σε αυτό το τομέα. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε τρόπου για να υπάρξουν περισσότεροι τέτοιοι εμπειρογνώμονε. Για παράδειγμα, η ανταλλαγή νέων αξιωματικών μέσω του στρατιωτικού Εράσμου αποτελεί μία από τις ε, εναλλακτικέ μας και οι στρατιωτικέ ακαδημίες θα πρέπει να προσφέρουν αντίστοιχη ε, εκπαίδευση. Επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα της ε, κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ευρείε τεχνολογικέ πλατφόρμες και να δημιουργήσουμε μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι μέσω μια τέτοια πλατφόρμα θα προβαίνουν σε περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και ασκήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται όλο ένα και περισσότερο και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Και ένας από τους τομείς συνεργασίας είναι η άμυνα στον κυβερνοχώρο. Μπορούμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συνεργασία, αλλά για να το επιτύχουμε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε νέες προτεραιότητες. Έχουμε καταρχήν το κέντρο αριστείας σε ό,τι αφορά ε, τη συνεργασία στον κυβερνοχώρο, όπως και το κέντρο αριστείας σε ό,τι αφορά την κυβερνοάμυνα ε, στο Ελσίνκι. Αλλά τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσουν την επιχειρησιακή του συνεργασία και το συντονισμό του, αλλά και να επιτείνουν τι ε, προσπάθειέ του για την αύξηση των ικανοτήτων. Οι ε, κοινέ δραστηριότητε κατάρτιση, η αύξηση, η δημιουργία περισσότερη εμπιστοσύνη και κοινέ ασκήσει ε, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για να επιτευχθεί αυτό. Επίση, θα πρέπει αυτό το περίπλοκο ζήτημα ε, να λάβει ε, υψηλότερη πολιτική προτεραιότητα. Άρα λοιπόν και το ε, φόρουμ που διοργανώθηκε το περασμένο φθινόπωρο του 2017 για τους Υπουργούς Άμυνας ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και ο ρόλος ο ηγετικός που ανέλαβαν οι δύο αυτές οργανώσεις είναι πολύ χρήσιμος για όλους. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό σε ό,τι αφορά την άμυνα στον κυβερνοχώρο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ αλλά και άλλων ε, εταίρων. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι το να εξετάσουμε πώς θα φτάσουμε σε μια κοινή συμφωνία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κοινών κανόνων και διατάξεων στον κυβερνοχώρο σε παγκόσμια κλίμακα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι παρότι η ομάδα κυβερνητικών Εμπειρογνωμών των ΗΕ δεν ήταν σε θέση να συντάξει μια έκθεση τη οποία συμφωνούσαν όλοι, η προηγούμενη έκθεση ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που ισχύει ε, ε, για όλους σε ό,τι αφορά ε, το κυβερνοχώρο. Το εγχειρίδιο του Ταλίν 2.0 αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση και εξηγεί το πώς μπορεί να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά το κυβερνοχώρο. Ωστόσο θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω κοινέ προσεγγίσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την κυβερνητική διπλωματία αλλά και την εφαρμογή ε, προτύπων βασικών κανόνων σε διμερές ε, επίπεδο σε ό,τι αφορά ε, δραστηριότητε στον κυβερνοχώρο. Τέλος, σε ό,τι αφορά την στρατιωτική και τη μη στρατιωτική συνεργασία, να πούμε ότι και εδώ πάλι η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι ζωτική σημασία. Θα πρέπει δηλαδή να αυξήσουμε και την εμπιστοσύνη ανάμεσα ε, και στις επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας και στους πολίτες. Θα πρέπει δηλαδή να επιτύχουμε ε, τη δημιουργία ενός ε, μιας κοινή αγοράς σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια. Χρειαζόμαστε ε, περισσότερη πρακτική υποστήριξη και απέναντι στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ακριβώς μπορούν να παρέχουν καινοτόμες λύσεις σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια. Και το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα ε, αλλά και άλλα ε, στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου μπορούν να παράξουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη. Άρα λοιπόν, ε, κλείνοντα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την πολιτική μα ό,τι αφορά την άμυνα στον χώρο Θα πρέπει να επιτείνουμε τη συνεργασία μα με τον ΝΑΤΟ και με άλλε χώρε που συμμερίζονται τι αξίε μα. Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερε κοινέ κατακτήσει και ασκήσει, αλλά και να αυξηθεί το accountability, δηλαδή η ανάληψη τη ευθύνη. Και αυτό γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουμε δει μέχρι σήμερα ε, και επειδή βέβαια ε, στο μέλλον οι σχετικές επιχειρήσεις πάντοτε θα περιλαμβάνουν όλο και περισσότερο αυτή τη διάσταση. Αυτά από την ε, πλευρά μου. Αναμένω τα σχόλια βέβαια από την πλευρά των υπόλοιπων στιγμών εισηγητών αλλά και τα σχόλια που θα ακουστούν στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ, ο κ. Λόπης White. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πάιτ για την έκθεση. Ποιοτική έκθεση. Και θα ήθελα να σχολιάσω κάποια σημεία. Κυρίως να επενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει πιο έντονη την προώθηση των προϊόντων ασφάλειας μέσω επενδύσεων, καινοτομίας, ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία στις αρχικές φάσεις της έρευνας και κοινοτομίας σε σχέση με την ασφάλεια στον κευνό χώρο σε διάφορους τομείς, υγεία, ενέργεια, χρηματοοικονομικά και βεβαίως άμυνα. Σήμερα μια ευρεία πλειοψηφία Ευρωπαίων πολιτών διαθέτει ίντερνετ που τελικά όπως ξέρουμε, ανέκυψε ως σύστημα επικοινωνίας που είχε αναπτυχθεί σε στρατιωτικό επίπεδο το 69. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πολιτικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του στρατού, όπως τα drones ας πούμε. Και επίσης και η αυτοματοποίηση μέσω της, ε, της μέσω των υπολογιστών. Έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις που θα πρέπει να προκαταλάβουμε. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια κοινή αγορά ασφάλεια στον κυβερνό χώρο που θα είναι καλά διαβαθμισμένη με τις καινοτομίε και που θα βοηθά τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να υπάρχει βιώσιμη και ταχύα ανάπτυξη. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αυτό προτείνει το κόμμα του ΕΛΚ, σε σχέση με την ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας πολιτικής και θεωρητικής σε αυτό το θέμα στην Ένωση, ώστε να προγραμματίσουμε ε, παρεμβάσεις γρήγορες και αποτελεσματικές. Θα πρέπει βεβαίω να πούμε ότι ο σχεδιασμός αυτός για την άμεση χώρο είναι καλό να προκαθοριστεί, γιατί θεωρώ ότι η ύπαρξη μιας ε, αρχής θα πρέπει να αποτελεί ένα είδος κέντρο επιχειρησιακού για όλες τις ε, χώρες μέλη, σε συνεργασία πάντοτε με τον ΝΑΤΟ, ώστε να είναι σε θέση να συντονίσει την ικανότητα αντίδραση στον χώρο μέσω σαφών παρεμβάσεων και κυβερνητικής δύναμης, μάλλον κυβερνοχωρητικής δύναμης, στα πλαίσια της κοινή πολιτικής αμήνας και ασφάλειας και στα πλαίσια επίσης της ΠΕΣΚΟ, του πλαίσιου μονιμής Αυτή η αρχή στον κυβερνοχώρο θα είναι αντικείμενο εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών και θα ακολουθεί βεβαίω και τι οδηγίε των Ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με θέματα πληροφοριών. Για να υποστηριχθεί αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα πρέπει βέβαια να έχουμε συμμετοχή υψηλόβαθμων βαθμών αξιωματικών εκ μέρου των χωρών μελών και κυρίω να υπάρχει συντονισμό με του υπουργού εξωτερικών και την ύπατη εκπρόσωπο. Η δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνα, όπω επιθυμούμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να ολοκληρώσουμε το τραγωνισμό του κύκλου, δηλαδή το άρθρο 42 τη της Λισαβόνα, Αυτό Αφορά δηλαδή τη δημιουργία μιας κοινή πολιτικής άμυνας μέσω μιας εναρμόνισης και διαφάνειας για όλες τις χώρες μέλη. Ένα Ευρωπαϊκό λοιπόν Συμβούλιο Άμυνας θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της, πολιτικής, πολιτική ε, στρατηγικής πολιτικής για την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή είναι ένα παγκόσμιο πεδίο χωρί σύνορα, θα πρέπει να, να γνωρίσουμε τι ικανότητέ μα και τι επιθετικέ και τι αμυντικέ στον κυβερνοχώρο, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο πολιτικό συντονισμό στην ε, διπλωματία στον κυβερνοχώρο και με τα απαραίτητα εργαλεία σε αυτό το πεδίο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσον αφορά την άμυνα στο κυβερνοχώρο θα έχουμε συνεχείς εξελίξεις και θα είναι όλο και πιο δύσκολο για τους νομοθέτες να προκαταβάλουμε τις εξελίξεις οι οποίες ε, παραμένουν άγνωστες. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να διαθέτουμε τους μηχανισμούς αναθεώρησης οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να εξυγχρονιστούμε σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την συνεργασία, ευχαριστώ και για τις τροπολογίες και τέλος, ε, Πρόεδρε, να με συγχωρήσετε γιατί θα πρέπει να φύγω αυτή τη στιγμή από την αίθουσα. Έχω καθυστερήσει, πάντως να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω για αυτό το ζήτημα που οπωσδήποτε θα είναι θέμα μεγάλη σημασία, όπω είπε και ο εισηγητή, και που βεβαίω υποστηρίζω για το μέλλον τη ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Λόπες. Τώρα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Μούντι, αντιπρόεδρος της ΕΔΕ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για ένα ήδη αξιόλογο σχέδιο έκθεσης, ε, καλά διαρθρωμένο, καλά συγκροτημένο, ε, που επισημαίνει τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και οι συνέπειες μιας κατάλληλης ε, άμυνας στον χώρο θα αγγίξουν κάθε πτυχή της ζωής μας σχεδόν, γιατί έχουμε ψηφιακά συνδεδεμένη τεχνολογία και από αυτή την άποψη μας καθιστά ευάλωτους. Οπότε είναι ευρωπαϊκή ευθύνη να θεσπίσει ποιοτική άμυνα στον κυβερνοχώρο. Αυτό απαιτούν ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης, είδαμε από κυβερνοεπιθέσεις ε, ότι μπορεί να είναι και στοχευμένες και είδαμε τις συνέπειες, αλλά μπορεί να είναι και προσπάσα κατεύθυνση. Γιατί είχαμε μια τέτοια ε, επίθεση στην Ουκρανία που προκάλεσε τεράστιες ε, ζημιές ε, σε επιχειρήσεις και οργανώσεις και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στη Ρωσία. Οπότε μπορεί να είναι ή στοχευμένες ή αδιάκριτες τέτοιες επιθέσεις. επίσης, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάποιους διεθνείς κανόνες και υπάρχει ε, τέτοια επιτακτική ανάγκη διεθνών κανόνων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αντίδρασή μας ε, στις κυβερναπιθέσεις. Και θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να εκλεπτύνουμε κάπως την έκθεση, συνεργασία με τον εισηγητή. Βέβαια θέλουμε κάποιες ικανότητες ε, κυβερνοάμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην δημιουργία εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Εκεί θα επιφέρουμε τη δική μας υπεραξία, προστιθέμενη αξία σε αυτό που γίνεται, όχι μόνο σε μεμονωμένες χώρες, αλλά σε συγκεκριμένα υπουργεία μεμονωμένων χωρών και να πρωτοστατήσουμε στο συντονισμό όλου αυτού του έργου που γίνεται μεμονωμένα, δημιουργώντας ένα μηχανισμό συνεργασίας και εμπιστοσύνης, ενισχυμένης συνεργασίας και ενισχυμένης εμπιστοσύνης. Η έκθεση επίσης ε, δίνει έμφαση στην ε, συνεργασία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΝΑΤΟ. Ε, και μάλιστα αυτός ο τομέας της κυβερνοάμυνα ήταν από του πιο επιτυχημένου ό,τι αφορά τη συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ. Και θα πρέπει και αυτή να ενισχυθεί όσο γίνεται. Επίση θα πρέπει μέσω των πολιτικών μας δικτύων να δίνουμε τις πληροφορίες στο ΝΑΤΟ για να αποφύγουμε επίθεση των στρατιωτικών δικτύων και θα πρέπει να γίνεται ταχεία μετάδοση, έως και αυτόματη μετάδοση των πληροφοριών. Επίσης, ένας άλλος τομέας πολύ σημαντικός είναι το θέμα της ανάθεσης. Γιατί ε, το Νοτπέτια στην Ουκρανία ε, ε, ίσως δρομολογήθηκε από κάποιους ρωσικούς κρατικούς φορείς, αλλά δεν υπάρχει μόνο το θέμα το κρατικό. Θα πρέπει να δούμε την αλυσίδα της κατά ανάθεση ανάθεσης και από αυτήν την άποψη η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη και έχει νόημα. Επίσης, δημιουργία ικανοτήτων, τεχνογνωσίας, έρευνα και τεχνολογικής ανάπτυξης που χρειάζεται σε ένα τομέα που έχει ραγδαίες εξελίξεις. Βέβαια, θα πρέπει να αντιληφθούμε την περιπροκότητα του θέματος. Δεν μιλούμε για παραδοσιακή κλασική άμυνα. Ξεπερνά την παραδοσιακή αντίληψη που έχουμε για την άμυνα και δεν είναι μόνο στρατιωτικό το σκέλος αυτής της άμυνας, έχει και πολιτικό σκέλος, γιατί έχουμε βαναπιθέσεις ε, στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, που επηρεάζουν τις υποδομές υγειονομικές, αλλά μπορούν να επηρεάσουν οποιοδήποτε άλλο τομέα. Και αυτό είπα στην αρχή. Ε, οι πολίτες μας ε, απαιτούν και εξαρτώνται από μας. Ε, γι' αυτό έχουμε καθήκον να αναπτύξουμε μια τέτοια πολιτική και θα συμβάλλω στην διαμόρφωση μιας καλύτερης έκθεσης. Πάντως χαίρω ήδη τον εισηγητή για το μέχρι τώρα έργο του. Εγώ είμαι και εισηγητρία των συντηρητικών μεταρρυθμιστών και πραγματικά επειδή ήταν εξαιρετικές οι παρατηρήσει των προελισάντων, δύσκολο είναι να προσθέσω τίποτα καινούριο. Θα ήθελα απλώ να σας υπενθυμίσω την προηγούμενη αποστολή μας ε, σε πολύ σημαντικά κέντρα. Στην Εστονία πήγαμε στο Τάλιν και εκεί επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κυβερνοάμυνας που είναι διαπιστευμένο από το ΝΑΤΟ στο Τάλιν και έγινε πολύ σημαντική ενημέρωση μια μάλιστα και από την Υπουργό Άμυνας της Εστονίας για το συγκεκριμένο αυτό κέντρο ε, και την ειδική ενημέρωση που έγινε προς υπουργού Άμυνας κατά την Ασθενική Προεδρία. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η ενημέρωση. Και καλό θα ήταν να, να ληφθεί υπόψη και από άλλους φορείς. Η ε, δεύτερη μας αποστολή έγινε στο Ελσίνκι στο Κέντρο Αντιμετώπιση Βρυδικών Απειλών ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Πάιτ θα επηρεάσει και τη σχετική έκθεση για το συγκεκριμένο κέντρο. Είναι πολύ χρήσιμη η πείρα της Εστονίας ε, στα θέματα κυβερνοάμυνας που είναι αρκετά προηγμένη, γιατί η Ιστονία ενέκυψε στο θέμα αυτό σχετικά νωρί. Είχαμε διάφορα περιστατικά επιθέσεων εις βάρος των υποδομών αυτής της χώρας και έτσι ευαισθητοποιήθηκε πολύ γρήγορα η χώρα αυτή στα ζητήματα των κυβερνοεπιθέσεων. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ του στρατητικού και του πολιτικού σκέλους στα θέματα της κυβερνάμινας. Να μην περιοριστούμε μόνο σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, γιατί η κυβερνοάμυνα έχει και πολιτικό σκέλος. Και εκεί υπάρχει λαμπρό πεδίο συνεργασίας και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και μάλιστα με τη μακροχρόνια πείρα του ΝΑΤΟ σε αμυντικά ζητήματα, σε συνδυασμό με τις δικές μας ικανότητες ε, και δεξιότητες και στα πολιτικά θέματα, πιστεύω ότι ε, θα κάνουμε τη διαφορά στη συνεργασία. Και μάλιστα το θέμα του κυβερνοχώρου αναφέρθηκε ως πρωταρχικός τομέας συνεργασίας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και μάλιστα προτάθηκαν και πιλωτικά προγράμματα και γυμνάσια, κοινέ ασκήσει για τη μετώπιση επιθέσεων. Αυτά και επαναλαμβάνω τα συγχαρητήριά μου προς τον συνάδελφο Ορμάς Πάιτ για την πολύ ισορροπημένη έκθεσή του, για το πολύ ισορροπημένο σχέδιο έκθεσης και που θα αποτελέσει πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση με τους και οδησηγητές και στην Επιτροπή και θα υποβληθούν φυσικά και συμβαστικές λύσεις. Ο Ίντρεκ Τάραντ τώρα, επίσης και οδησηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το σχέδιο έκθεσής του και να το κάνω κρυπτογραφημένα σε μια γλώσσα κρυπτογράφησης που ο κύριος ε, Πάετ την κατέχει. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία αυτή θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των αμυντικών μας κονδυλίων και ότι τα θέματα, ο της ασφάλειας και της άμυνας αυξάνεται και ευτυχώς, γιατί έχουμε και μία οικονομική ανάκαμψη και μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε υψηλότερο προπολογισμό. Όμω ε, τα κονδύλια μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ασφάλεια και άμυνα ε, σε σύγκριση με τα αμερικανικά ε, υπολείπονται. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη μελέτη του Τμήματο Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδειξε ότι οι αμυντικέ δαπάνε των ΗΠΑ είναι πολύ πιο αποτελεσματικέ από τι αντίστοιχε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιάνουν καλύτερα τόπο τα κονδύλια μας σε θέματα αυτά δημιουργίας αμυντικών ικανοτήτων. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες ε, διευκρινήσεις ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή και τον ορισμό του όρου κυβερνοάμυνα ή άμυνα στον κυβερνοχώρο. Γιατί μπορεί να εξεταστεί είτε ε, διασταλτικά είτε συσταλτικά αυτή η έννοια. Καταρχήν, ποιον θέλουμε να προστατεύσουμε από τις ε, κυβερνοεπιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις και οι στρατικές δομές καλύπτονται από την παράγραφο 28. Ο κύριος Πάετ αναφέρθηκε και στην προστασία των πολιτικών υποδομών. Περιλαμβάνουμε και κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές ή μόνο υποδομές που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ε, την προστασία και την υγεία. Ή μήπω μιλάτε για υποδομέ που έχουν ε, κέριο, ε, κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της οικονομίας. Θα πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε ε, θέλει να προστατεύσει και επίση τι είδου κακόβουλες απειλέ θέλουμε να αποτρέψουμε. Γιατί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ε, πολιτική, οικονομική στόχη, ε, το η κυβερνοκατασκοπία, η προπαγάνδα, η fake news, η πρόσβαση, περιορισμένη πρόσβαση στο ίντερνετ, τι είδους κακόβουλες επιχειρήσεις θέλουμε να αποτρέψουμε. Οπότε και το πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να καθορίσουμε, γιατί άλλη προσέγγιση έχουμε με την ε, προστασία κρίσιμων υποδομών και άλλη με την προστασία από φαλκιδευμένες ειδήσει ή από ψευδή ενημερωτική προπαγάνδα. Επίσης, είχαμε ένα σκάνδαλο με μια ε, επιχείρηση, την Cambridge Analytica. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τους πολίτες από κάποιες εταιρείες, ε, κάποιες εταιρείες όπως την Cambridge Analytica που προσπάθησε να ε, παραπλανήσει ή να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών. Ερήμην ε, κυρία Φωτίγα, εσείς του χρόνου θα αντικατασταθείτε από ε, εταιρείες σαν την Cambridge Analytica. Θα πρέπει να προασπίσουμε και τη δική σας θέση και το δικό σας θόκο. Και τέλος, πάλι για το πεδίο εφαρμογής. Ποια είναι η επίσημη εντολή και μπορεί να είναι βαρετό το θέμα και κουραστικό, αλλά ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάποια συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών που διεκδικούν την κατουσία αρμοδιότητα για την έκθεση. Στα τέλη του 2017 είχαμε ε, μια σύγκρουση μεταξύ των επιτροπών ΙΜΚΟ και σε ό,τι αφορά την εντολή της έκθεσης ΠΑΕΤ. Και η ΙΤΡΕ είχε έκθεση πρωτοβουλίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την οποία διεκδίκησε η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτού. Οπότε θα ήθελα να, πω, να ρωτήσω τον κύριο Συγητή να μου πει πώς ε, επιλύθηκε τελικά, πώς διαθετήθηκε αυτή η διαφορά και η αφισβήτηση, η σύγκρουση αρμοδιότητα μεταξύ των τριών επιτροπών και πώς θα αποφύγουμε επικαλύψη με τις άλλες δύο επιτροπές, ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ, στην ε, υποεπιτροπή μας. Εγώ δεν είμαι μέλος ούτε της ΙΤΡΕ ούτε της ΙΜΚΟ, γι' αυτό θα υποστηρίξω τα δικά μας ε, προνόμια και αρμοδιότητες της ΕΝΤΕ. Ναι, ε, να, απλώς να επιβεβαιώσω ότι ε, προφανώς ισχύει αυτό ότι το μέλος της κάθε επιτροπής προσπαθεί να προωθήσει τις αυτής της επιτροπής. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σκανδαλό, απλώς τα όσα συμβαίνουν, τα γεγονότα δηλαδή, ο αριθμός τους ε, υπερβαίνει ε, τις ε, οργανωτικές δυνατότητες οποιοδήποτε θεσμικού οργάνου. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο και της διάσκεψης των Πρόεδρων των Επιτροπών. Υπάρχει και από εκεί και μετά βέβαια και μια διαδικασία διαιτησίας και ούτω καθεξής. Ο κύριος Μπόγκταν Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι μου αρέσει πολύ η έκθεση ΠΑΕΤ. Θεωρώ ότι είναι ε, μεστή, ισορροπημένη σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής. Αλλά κατά τη γνώμη μου Ε, φαίνεται ότι ο εισηγητής της ε, έκθεσης είναι ένας πολύπυρος διπλωμάτης. Ε, για παράδειγμα, μόνο δύο φορές σε ολόκληρη την έκθεση αναφέρεται το απαιτεί. Τέσσερις φορές στην έκθεση αναφέρεται το απευθύνει έκκληση πολύ περισσότερο αναφέρει το με ικανοποίηση σημειώνει. Είναι πάρα πολύ διπλωματική διατύπωση της έκθεσης, οπότε ίσως δώσουμε την εντύπωση ότι στα θέματα του κυβερνοχώρου έχουμε μια κατάσταση που μπορεί να μην ελέγχουμε πλήρως, αλλά σίγουρα ακολουθεί μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Αλλά όταν διαβάζουμε την έκθεση, όλα αυτά τα θέματα που περιλαμβάνονται δείχνουν μια, κάποιες ελλείψεις. Δεν έχουμε πυρογνώμονες, έχουμε κενά στην εκπαίδευση, δεν έχουμε τεχνικές πλατφόρμες, έχουμε χαμηλό επίπεδο λήψης αποφάσεων σε θέματα κυβερνοχώρου, έχουμε νομικά κενά σε όλα τα επίπεδα και σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε κατακαιρματισμό αρμοδιοτήτων, υπερβολικά αργή αντίδραση σε ραγδαίες εξελίξεις. Οπότε στην ουσία είναι πολύ επικριτική η διατύπωση, η έκθεση, αλλά η διατύπωση παρά είναι διπλωματική και δίνει κάπως διαφορετική ιδέα. Και έχουμε μια αίσθηση, αν όχι σχιζοφρένειας, μεταξύ διατύπωσης και ουσίας, αλλά ε, μιας διαφοράς. Οπότε αν δεν έχουμε μια πιο ισχυρή διατύπωση, ίσως δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, ενώ το αντίθετο ε, δείχνει η έκθεση. Οπότε, ναι μεν περιλαμβάνεται ουσιώδη ουσιώδη έκθεση, αλλά η διατύπωση είναι υπερβολικά διπλωματική και χαλαρή. Οπότε, μερικές εκφράσει εκφράσεις ικανοποίηση να τις αντικαταστήσετε από μια πιο απαιτητική διατύπωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άρνε Λίτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Speak English. Um, Θα μιλήσω στα αγγλικά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχέδιο έκθεσης, ε, στο οποίο ε, θίγεται μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα ε, σε ό,τι αφορά και την κυβερνοεπίθεση στη Γερμανία. Νομίζουμε πως είναι από τη Ρωσία και αυτό που αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ίσως θα μπορούσαμε εδώ να αναγνωρίσουμε ε, με κάποιο τρόπο τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες των κρατών γιατί τελικά σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Για παράδειγμα, όταν ε, ε έρχομαι σε επαφή με έναν συνάδελφο από το ΕΣΠΕΤΗ που είναι αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα, μου λέει ότι δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά. Ε, περισσότερες δηλαδή αρμοδιότητα ε, τη Ένωσης ε, εδώ. Και θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και μεταξύ μας εδώ ω προ το τι θέλουμε. Από εκεί και μετά νομίζω πως ε, και μετά από αυτήν την κυβερνοεπίθεση αλλά και άλλε επιθέσει ανά τον κόσμο χρειαζόμαστε ένα διεθνές δίκαιο για τον κυβερνοχώρο. Θα χρειαστούμε δηλαδή ψηφίσματα στο μέλλον των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις που λαμβάνουν χώρα όπως υπήρξαν και ψηφίσματα για παράδειγμα της Ένωση ό,τι αφορά το φυσικό αέριο ή άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν, ενδεχομένω, παρότι βέβαια πρόκειται για έκθεση της ΕΣΕΝΤΕ, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιε προσπάθειε να ξεκινήσει δηλαδή μια διαδικασία ούτως ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στην επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή ενό διεθνού δικαίου για τον ε, ε, χώρο. Ίσως δηλαδή να πούμε ότι τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνουν μια αναφορά, για παράδειγμα τα κράτη-μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω σε ό,τι αφορά το Brexit, ότι η κυρία Τερίζα Μέη ε, πήγε και σε μια ε, διάσκεψη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και αυτό το ζήτημα αφορά βέβαια όχι μόνο τους τρόλους για παράδειγμα στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά αφορά και γενικότερα τις ικανότητες σε αυτό το τομέα. Έχουμε τα όσα γνωρίζουμε σε σχέση με τη Ρωσία αλλά από εκεί και μετά ε, θα πρέπει να δούμε και στο μέλλον πώς ε, θα εξελιχθούν τα πράγματα με την Κίνα η οποία αυξάνει πάρα πολύ τις ικανότητες της εδώ και αναφέρθηκε επανειλημμένα σε αυτή τη διάσκεψη η Κίνα. Ε, η κυρία Τερίζα με ανέφερε σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι προς το συμφέρον και της Μεγάλης Βρετανίας να συνεχίσει να συνεργάζεται σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. με οποιαδήποτε και αν είναι παρέμβαση, για παράδειγμα όπως αυτή που αναφέρατε, διάλογος δηλαδή και με την ε, Νέα Ζηλανδία και με την Αυστραλία ή με τις άλλες χώρες όπως με την Μεγάλη Βρετανία, είναι πάντοτε σημαντικό να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να βασιζόμαστε ε, στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και μετά εμείς. Και στο πλαίσιο του μελλοντικού διαλόγου που θα γίνει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, νομίζω πως θα πρέπει να εξετάσουμε ακριβώς την ε, κοινή πολιτική κύβερνο ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου και τα κράτη-μέλη να ενοποιήσουν, να εναρμονίσουν περισσότερο τις ε, πολιτικές τους ε, στον κυβερνοχώρο. Για να υπάρξει μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή διαστάση σε σχέση με αυτό το ζήτημα και να υπάρξει περισσότερη έρευνα σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω με ενδιαφέρον τις τη μελλοντική μας συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Λίτς. Και σίγουρα α, θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ε, μία σειρά από τα σημεία τα οποία αναφέρατε στις ε, επόμενες συνεδριάσεις ε, που θα γίνουν στη ΣΕΔΕ αλλά και σε συνεργασία με άλλες ε, επιτροπές ε, καθώς ε, πρόκειται για ζητήματα τα οποία άπτονται εδώ τόσο εθνικής όσο και διεθνούς νομοθεσίας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά και το ζήτημα δυνητικών μελλοντικών κυβερνοεπιθέσεων, τις οποίες είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πού προέρχονται. Ο κύριο Κάρβερ έχει τώρα το λόγο και συνέχεια ο κύριο Εποστινάδου. Ναι. Ε, μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Ε, μετά από τα όσα είπε ο κύριο Λίτζε σε ό,τι αφορά δηλαδή, τα ώρα που θα πρέπει να θέσουμε, νομίζω πω ε, σε μια συνεδρίαση τη ΑΦΕΤ είχε γίνει μια συζήτηση πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit και γνωρίζετε ποια είναι η θέση μου σχέση με εκείνο το δημοψήφισμα. Ε, εγώ θεωρούσα ανέκαθεν ότι είναι προ όφελο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία με, το, ε, με, με τη Μεγάλη Βρετανία και πολλέ από τι ιδιαίτερε πληροφορίε που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από εκεί. Οπότε, ακόμα και αν εγκαταλείψει πραγματικά η, η Μεγάλη Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστεί να συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ μα. Ε, και να δούμε και τι θα γίνει και στο επίπεδο γενικότερα της πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας. Πάντως η συνεργασία στον ε, κυβερνό τομέα είναι σίγουρα απαραίτητη ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, δεν είναι μόνο έγκαιρη και κέρια έκθεση, αλλά απαραίτητη γιατί αυτή η απειλή είναι μια από τις πιο ευρείες και πιο διστραμμένες απειλές, γιατί έστω και αν κάνουμε ένα ακριβή ορισμό της κυβερνοεπίθεσης και του κυβερνοπολέμου, θα δούμε ότι είναι δύσκολο να καθορίσουμε και να διαχωρίσουμε τι είναι πολιτικό και τι στρατιωτικό. Συνήθως στις κυριότερες οι μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις έχουμε και στις δύο πλευρές, πολιτικές και στρατιωτικές ή πολιτικές με σοβαρές στρατιωτικές επιπτώσεις. Γι' αυτό ακριβώ είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τι είναι καθαρά στρατιωτικό, αμυντικό και τι πολιτικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα σε ένα ψηφιοποιημένο κόσμο και οικονομία με την ε, πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν απειλή, ενδεχόμενη απειλή. Επειδή όσο προχωράμε στην δικασία ψηφιοποίησης, τόσο περισσότερο εξαρτώμαστε από τη τεχνητή νοημοσύνη και τόσο πιο ευάλωτοι είμαστε. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό η Ευρώπη επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της και να επενδύσει στην έρευνα και στην ανάπτυξη ώστε να αναπτυξεί την τωρινή της δυνατότητα εντοπισμού των απειλών να αμυνθεί από τις τρέχουσες ε, επιθέσεις και ενδεχομένω να απαντήσει. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται ανησυχητικό ή επιθετικό, αλλά αν κυρίως είσαστε μόνο καλοί και παρακαλάτε και τέβετε τους άλλους μή το κάνετε, σας παρακαλώ σταματήστε τις επιθέσεις, τότε αν δεν έχετε την αξιόπιστη δυνατότητα απάντησης, τότε χαθήκαμε. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και να επενδύσουμε αυτή τη δυνατότητα ανταπόκρισης, απάντησης. Νομίζω σε, σε αυτές τις καταστάσεις κανείς δεν γλιτώνει. Κανείς δεν γλιτώνει από τις κυβερνοεπιθέσεις. Είχαμε μια μεγάλη ε, κυβερνοεπίθεση ε, στις Πολιτείες, στην ε, υποδομή ενέργειας, με τεράστιους, με κολοσσούς επιχειρήσεις, με προηγμένα συστήματα άμυνας. Παρ' όλα αυτά ήταν στόχος και στη ΣΥΠΑ λοιπόν, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τις καλύτερα προετοιμασμένες ε, χώρες στον κόσμο, δέχτηκαν κυβερνοεπιθέσεις. Γερμανία, δύο σημαντικά υπουργεία δέχτηκαν σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τις λεπτομέρειε της καταλανικής κρίσης και θα δούμε και εκεί πτυχές κυβερνοεπίθεσης υβριδικής κατά των ισπανικών συμφερόντων. Για μιλήσω και για τις μικρότερες χώρες όπου μάλιστα οι πιο μεγάλες πολιτικές, συγγνώμη, στρατιωτικές δυνάμεις και οι καλύτερα εξοπλισμένες ε, στρατιωτικές χώρες αν αυτές είναι ευάλωτέ, τότε πώς μπορούμε να διανοηθούμε ότι οι μικρές χώρες θα μπορέσουν να αμυνθούν. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επιμείνουμε ότι μόνο μια ικανότητα απάντησης ευρωπαϊκή μπορεί να μας βοηθήσει να προστατευτούμε και να αμυνθούμε ώστε μελλοντικά να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιους κινδύνους. Και μια τελευταία παρατήρηση. Πιστεύω ότι σε αυτή την οργουελική κατάσταση θα πρέπει να δούμε το συσχετισμό των διαφόρων προσεγγίσεων μας. Δηλαδή, πώς θα προετοιμάσουμε τις οικονομίες μας, πώς θα προετοιμάσουμε τις κοινωνίες μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιθέσεις. Πώς μπορούμε εν τέλει να προετοιμαστούμε εμείς οι ίδιοι ώστε νομικά να προσδιορίσουμε οι ελευθερίες και τα δικαιώματα που προστατεύονται και που υπό απειλή, οι απειλούμενοι θα πρέπει να επιτρέψουμε τη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και να καταλήξω με τα FEE e, αυτοκίνητα, FEE e πόλεις που διαθέτουμε κτλ. κτλ. Όλα αυτά όσο πιο FEE e γίνονται, τόσο πιο ευάλωτα γίνονται. Και σήμερα το πρωί διάβασα ότι ένα παλιό σοβιετικού τύπου κινέζικο τάγκ μετατρέπεται σε FES τάγκ με τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει σε αυτό το παλιό τάγκ της δεκαετίας του 50 να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα τα οποία είναι εξοπλισμένα με στατικό εξοπλισμό τεχνικής ε, νοημοσύνης, δηλαδή ντρόν, δορυφόροι κτλ. Ένα παλιό τάκ του 50, έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα και θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς, γιατί η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα και αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στον τοίχο των δακρύων και να διαμαρτυρόμαστε, τότε θα χαθούμε και πραγματικά η Ευρώπη για διάφορους λόγους αποτελεί στόχο άλλων παγκοσμίων δυνάμεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ θερμά. Και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν σε θέση να παρακολουθήσω την παρουσίαση του κύριου Πάτ. Αλλά υποστηρίζω τα όσα περιλαμβάνει το σχέδιο εκθεσής του. Όμως η παρέμβαση του κυρίου Μποστινάρου μου έδωσε το ένασμα το να επιχειρηματολογήσω ε, στις ίδιες ε, γραμμές ε, με αυτές που έκανε την παρέμβαση του μόλις τώρα. Δηλαδή αναφέρθηκε στη Γερμανία και στο γεγονός ότι βρέθηκε θύμα και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας επί σειρά μηνών ε, μια τέτοια κυβερνοεπίθεση. Ε, μεταξύ άλλων και το Think Tank ε, Ευρωπαϊκή Εταιρεία για Εξωτερική Πολιτική. Εκεί βλέπουμε πως υπεκλάβησαν κάποια έγγραφα σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και την Κίνα. Οπότε ακριβώς με βάση αυτήν την κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε τώρα μία πιο έντονη συζήτηση στη Γερμανία, όχι μόνο ως προς την άμυνα, αλλά ως προς και το πώς μπορούμε να ε, πιο ενεργοί. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε θύματα μιας επίθεσης, ε, να μπορέσουμε να αντεπιτεθούμε σε εκείνους ε, που μας επιτίθενται. Δηλαδή, η βασική μας θέση είναι ότι είμαστε φίλοι ειρηνικοί αλλά όταν βρισκόμαστε θύματα μιας επίθεσης δεν θα πρέπει απλώς και μόνο να προσπαθούμε να αμυνθούμε. Σε τεχνικό επίπεδο θα πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγικές οι οποίες θα μας επιτρέψουν, για παράδειγμα, να ε, προκαλέσουμε μια ζημιά, για παράδειγμα, στη συσκευή η οποία είναι υπεύθυνη για αυτήν την κυβερνοεπίθεση. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταφέρνουμε πολλά μόνο με άμυνα. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια πολύ δημιουργική συζήτηση ως προς το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού ως Ευρωπαίοι σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόντ. Äh, ευχαριστώ, θα μιλήσω στα γερμανικά. Αφού μίλησε και μόλις τώρα ο συνάδελφος Γκάλερ στα γερμανικά, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο έθεσε ο συνάδελφος εμποστινάρου και το οποίο έχει συζητηθεί μέχρι στιγμή κάπως ε, θεωρητικά, αλλά το οποίο θα μπορούσε να είχε πολύ πρακτικές συνέπειες ε, για όλους μας. Και εδώ αναφέρομαι σε κυβερνότητες, ε, σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, δηλαδή για παράδειγμα εργοστάσια παραγωγή ενέργειας. Εντάξει μπορεί κανείς να εξετάσει το, για παράδειγμα τι θα συμβεί αν σταματήσουν οι λειτουργίες, ε, για παράδειγμα μια εγκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ε, γνωρίζετε το τι θα σήμαινε αν σταματούσε η παραγωγή ενέργειας, ε, για παράδειγμα, σε μια χώρα. Ε, είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από την ε, ενέργεια σήμερα. γιατί δεν είναι ότι δεν θα λειτουργεί μόνο το ασατσέρ, για παράδειγμα. Δεν θα υπάρχει ούτε ίδρυυση, τροδότηση, δεν θα υπάρχει ούτε βενζίνη, δεν θα υπάρχει τρόπος να διαφύγουμε, εκτός κι αν είναι γεμάτο το δεπόζιτο του αυτοκινήτου, δεν θα υπάρχει, ε, δεν θα υπάρχουν άλλα ε, οπότε όλα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα της ε, ηλεκτρικής ενέργειας και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την προστασία των σχετικών υποδομών. Θα πρέπει δηλαδή να λάβουμε ιδιαίτερα μέτρα σε ό,τι αφορά την προστασία αυτών των υποδομών. Εντάξει, δεν είμαι ειδικό σε αυτά τα ζητήματα, αλλά νομίζω πως αυτή οι μεγάλη φορείς ε, ηλεκτρικής ενέργειας να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το διαδίκτυο και το ξαναλέω δεν είμαι εμπειρογνώμονας ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό. Δηλαδή, ίσω θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αποκοπεί, αν θέλετε, η τόσο μεγάλη σύνδεσή του με τον έξω κόσμο, έτσι ώστε να μην είναι εύκολο ακριβώ να βρεθούν θύμα μια επίθεση. Ε, Πρόεδρο, ε, συνάδελφοι, θα πρέπει να κλείσω εδώ το κατάλογο των ομιλητών, ε, γιατί πραγματικά έχουμε καθυστερήσει λίγο. Κ. Μποστινά, ζητάτε λόγο για μία πρόταση. Ναι, συνήθως εκείνοι οι οποίοι προβαίνουν σε κύβρονο είναι είτε κρατικές, κρατικοί φορείς, είτε ε, κάποιες ομάδες ε, πάρα πολύ ε, μικρού μεγέθους. Οπότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε μία αντίδραση απέναντι στο μέγεθος εκείνο που προβαίνει σε κυβερνό επίθεση. Είναι δύσκολο να εντοπίζουμε ε, τον, ε, το ποιο έχει προβεί σε μία κυβερνό επίθεση γιατί διαφέρουν πολύ σε μέγεθος αλλά και επειδή μπορούν να μετακινούνται από ένα σημείο σε άλλο ε, πολύ γρήγορα. Πρόεδρος, ε, πρωτού ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Πάετ, ε, να σας υπενθυμίσω ότι 10 Απριλίου, έως τις 10 Απριλίου μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας, οπότε έχουμε σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Από εκεί και μετά θα υπάρχει μια δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης στις 15 Μαΐου, εδώ στις 11 και 16 Μαΐου 16 ή 17 λέει ο πρόεδρο, θα γίνει ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ. Εάν θέλουμε πράγματι να ψηφιστεί αυτή η έκθεση τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Άρα λοιπόν λάβετε υπόψη σας, σας παρακαλώ αυτούς τους χρονικούς ε, περιορισμούς. Ε, να ξαναδώσω τώρα το λόγο στον συγκεκριτή ο κύριος ε, Πάετ, αλλά λέγοντάς το ότι δεν μας μένει πολύς χρόνος. Ευχαριστώ πολύ συναδελφοί για τις ε, ιδέες σας, τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας και νομίζω πως ένα συμπέρασμα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχει πλέον περισσότερη συνείδηση σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα από τους ε, αρμόδιους για τη χάραξη τους, ε, της πολιτικής, τους ηθήνοντες. Και γνωρίζουμε ότι ναι, η αρμοδιότητα και για τη λήψη αποφάσεων βρίσκεται στα κράτη-μέλη, αλλά δεν ε, βρίσκεται και συντονισμό και συνεργασία μεταξύ του εκεί που θα έπρεπε σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική απόκριση τέτοιων επιθέσεων, ειδικότερα καθώ τέτοιου είδου επιθέσει μπορούν να έχουν θανάσιμε επιπτώσει. Τώρα, όπω έθεσε και ένα σχετικό ερώτημα ο συνάδελφο από του ε, Πρασίνου ε, σε σχέση με τα σχετικά όλα που θα βάλουμε, νομίζω πως με βάση τη συζήτηση που έγινε και πέρσι, αποφασίσαμε ότι θα εστιάσουμε σε αυτή την έκθεση κυρίως σε ζητήματα άμυνας, κυβέρνο άμυνας. Οπότε αντιλαμβάνομαι τις κοινέ που έχουμε εδώ αλλά ε, από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, διαχωριστεί ακριβώς η άμυνα από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δηλαδή τα στρατιωτικού και τα μη στρατιωτικού χαρακτήρα ζητήματα. Πάντως θα προσπαθήσω εδώ να λάβω υπόψη μου χρήσιμες και ουσιαστικές ε, τροπολογίες έτσι ώστε να βελτιώσουμε το κείμενο της έκθεσης Ευχαριστώ και για το σχόλιο που έγινε ότι σε ορισμένα σημεία είναι υπερβολικά διπλωματική η διατύπωση του σχεδίου της έκθεσης. Ίσως θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο εμφαντικό. Αλλά πράγματι βέβαια προσπαθούμε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ζητημάτων που θίγονται εδώ. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για τα σχόλιά σας και θα σας ξαναδώ τους και ότι όταν θα συζητήσουμε τις σχετικές τροπολογίες. Και βέβαια θα έχουμε και την δεύτερη εξέταση αυτού του σχεδίου το Μάιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Πάρτ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Τη σημερινή διάταξη, αλλά το επόμενο είναι συναφές με το προηγούμενο. Γι' αυτό παραμένετε παρακαλώ στην αίθουσα. Ε, θα γίνει παρουσίαση ενός πολύ καινοτόμου σχεδίου στα πλαίσια της μόνιμης διαρθρωμένη συνεργασίας και θα ήθελα να καλέσω το μόνιμο εκπρόσωπο της Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μας παρουσιάσει αυτό το καινοτόμο σχέδιο της ΠΕΣΚΟ για τις ε, ομάδες ταχείας αντίδρασης σε θέματα του κυβερνοχώρου. μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Μαρτζίρης Αμπουκεβίτσιους, Καλώς ήρθατε κύριε Μποκεβίτσιους στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής ΕΝΤΕ. Είστε επικεφαλής της ομάδας άμυνας της μόνιμης αντιπροσωπείας της Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μας κάνετε την παρουσίαση αυτού του καινοτόμου, όπως είπα, σχεδίου της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας τη σύσταση ομάδων ταχεία αντίδραση σε θέματα στον χώρο που έγινε με πρωτοβουλία τη Λιθουανία. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω και να σα παρουσιάσω αυτή την πρόταση. Καταρχήν, να κάνω λίγα σύντομα σχόλια που μου ήρθαν στο μυαλό από την προηγούμενη συζήτηση και να σας διαβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης, γιατί αυτό που επιδιώκουμε με το δικό μας σχέδιο του, της ΠΕΣΚΟ ε, είναι αυτό που ζητήσατε κι εσείς, δηλαδή αναβάθμιση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη συνεργασία του στρατιωτικού και του πολιτικού σκέλους και να μην περιοριστούμε στη δημιουργία κάποιου ανθεκτικότητας, αλλά να υιοθετήσουμε μια πιο προορατική προσέγγιση στις κυβερνοεπιθέσεις και στις κυβερνοαπειλές. Οπότε σας διαβεβαιώ ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και συμπνέουμε πλήρως τα θέματα αυτά. Καταρχήν ως προς το υπόβαθρο. Γιατί η Λιθουανία πρότεινε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η πρόεδρος διακόπτη. Λίγη ησυχία παρακαλώ στην αίθουσα, γιατί αυτή η φασαρία που ακούγεται ενοχλεί τον ομιλητή μας. Γιατί λοιπόν η Λιθουανία υπέβαλε τη σχετική πρόταση. Ε, το θέμα αυτό σχετίζεται με την ε, γενική στρατηγική που ε, δίνει τρία καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαχείριση κρίση για δημιουργία ικανοτήτων και προστασία τη Ευρώπη. Καταρχήν, διαχείριση των κρίσεων. Αυτό που κάνει συνήθω η Ευρωπαϊκή Ένωση στι ε, στρατιωτικέ επιχειρήσει και αποστολέ τη. Ε, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων. Έχει κάποιε σχετικέ δραστηριότητε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να τι εντατικοποιήσει. Και το τρίτο νέο καθήκον είναι η προστασία τη Ευρώπη. Και το βλέπουμε αυτό κυρίως στην προσπάθεια συμπλήρωσης του ΝΑΤΟ, γιατί η, το ΝΑΤΟ αφορά την άμυνα της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση την προστασία της Ευρώπης. Και προσπαθώντας να δώσουμε ένα νόημα σε αυτό το καθήκον στην προστασία της Ευρώπης, νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την προστασία από τις κυβερνοεπιθέσεις και την αποτροπή των κυβερνοαπειλών. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε και τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, την ΠΕΣΚΟ ε, διαβάζοντας τη συνθήκη της Λισαβόνας που περιέχει τις διατάξεις για την ΠΕΣΚΟ, διαπιστώνουμε ότι αφορούν περισσότερο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ε, επιχειρήσεων ασφάλειας. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε η ΠΕΣΚΟ να αντιμετωπίσει και τις ε, τρέχουσες απειλές. Και μάλιστα όταν συζητήσαμε τις δεσμεύσεις της ΠΕΣΚΟ, καταλήξαμε σε 20. Μία από αυτές είναι η ενίσχυση της ε, συνεργασίας σε θέματα ε, Άμυνα. Και μάλιστα συμπεριλάβαμε αυτή τη δέσμευση στον κατάλογο των καθηκόντων της ΠΕΣΚΟ. Και γι' αυτό θέλουμε να προτείνουμε συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ε, είναι πολύ ευαίσθητος ο τομέας αυτός, χρειάζεται οπωσδήποτε εμπιστοσύνη και να αρχίσουμε να σφυριλατούμε αυτή την εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι αντιλαμβανόμαστε πως ε, καταρχήν ε, σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως και εκ παραλλήλου θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύοντας τη συνεργασία μας σε στα θέματα αυτά. Η ΠΕΣΚΟ λοιπόν, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία είναι το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο γιατί μιλά για τις αμοιβέ μας υποχρεώσεις και εξωθεί τα κράτη-μέλη να διευρύνουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα κυβερνοχώρου και ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Όπως είπα, η πρώτη αντιμετώπιση θα γίνει σε εθνικό επίπεδο και φυσικά συνειδητοποιούμε την ανάγκη, δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε την εθνική δημιουργία ικανοτήτων. Αλλά κάποια στιγμή καλό θα ήταν να αναπτύξουμε και ευρωπαϊκές ικανότητες που θα ενισχύσουν τις εθνικές ικανότητες. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας κάτι τέτοιο. Γιατί δεν αποκλείεται ακόμη και πολύ προηγμένες χώρες στα θέματα αυτά, όπως ακούσαμε παραδείγματα πριν στη συζήτηση, θα μπορούσαν κάλλιστα να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπου δεν αρκούν οι εθνικές αντιδράσεις, η εθνική αντιμετώπιση. Και εδώ δημιουργείται μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει τέτοιες ε, υπερεθνικές ικανότητες. Θα πρέπει βέβαια να υπερτιμούμε τη συγκεκριμένη πρόταση, το συγκεκριμένο project. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα πιλωτικό σχέδιο που θα δοκιμάσει διάφορες έννοιες και προτάσεις. Μία από αυτές είναι η αμοιβαία ε, συνδρομή στις ομάδες ταχείας αντίδρασης ε, στον κυβερνοχώρο. Δεν έχουμε αντλήσει ακόμη πολλά διδάγματα γιατί προσκουρέσαμε σε πολλές επιφυλάξεις Μερικοί δεν το θεωρούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τις κυβερνοαπειλές. Και όσοι δεν ξέρουν τα δίκτυα, δύσκολο είναι να το αντιληφθούν. Πάντως έχουμε μερικά πολύ θετικά παραδείγματα τέτοιας συνδρομής αμοιβαία. Και θέλουμε να αποδείξουμε την λειτουργικότητα αυτού του μοντέλου. Επίσης, άλλο τομέα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους. Βέβαια, η κυβερνοασφάλεια είναι εξορισμού διτή και στρατιωτική και πολιτική. Και υπάρχει έντονο πολιτικό σκέλος. αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους και νικτές δράσεις, στρατιωτικές και πολιτικές. Και αυτό μπορεί και από την ε, εθνική μας εμπειρία. Βέβαια κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα, αλλά εμείς στη Λιθουανία πρόσφατα ε, δημιουργήσαμε μια ενιαία ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική. Ένα τέτοιο ενίο κέντρο ΣΕΡΤ, όπως το λέμε, που είναι αρμόδιο για όλους τους κλάδου του τομεί. και για τον κυβερνητικό τομέα, και για το στρατιωτικό και για το πολιτικό. Ένα ενίο τέτοιο κέντρο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην πληροφορική πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλη έγκυση και θα ρίνουμε και τα άλλα κρατημέλη να μα μιμηθούν. Όπω είπα, το σχέδιο αυτό είναι πιλωτικό, είναι πειραματικό. Και θα έχει ένα προοδευτικό χαρακτήρα. Σε μία πρώτη φάση και με τις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα κάνουμε πρώτα μία νομική ανάλυση της κατάστασης, γιατί όπως είπα το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και το νομικό πλαίσιο δεν είναι και πολύ πρόσφορο για την παροχή ή την ε, αποδοχή συνδρομής από άλλες χώρες ακόμη και αν είναι κοινοτικέ. Οπότε στόχος μας είναι να κάνουμε μια περιεκτική διεξοδική νομική ανάλυση για το τι επιτρέπεται σε ό,τι αφορά τη συνδρομή των άλλων χωρομελών, τη συνδρομή κοινοτικών θεσμικών οργάνων και τι, τι είναι εφικτό σε ό,τι αφορά τη συνδρομή των εταίρων μας. Δεν μας φοβίζει μια απάντηση ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι όλα εφικτά ή δεν επιτρέπονται όλα. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να αλλάξει σε εθνικό επίπεδο, στην εθνική νομοθεσία. Επίσης, θέλουμε στις ομάδες μας αυτές να έχουμε κοινά γυμνάσια, κοινέ ασκήσεις. Η πρώτη κοινή άσκηση θα γίνει στα τέλη του τρέχοντος έτους. Το αισιόδοξο σενάριο είναι να έχουμε ήδη σε εφεδρεία μια ομάδα από τις αρχές του επόμενου έτους. Σε επιφυλακή. Να είναι ήδη έτοιμη. Και εδώ θα πρέπει να δώσω αρκετές εξηγήσει γιατί μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά οι συνάδελφοι τι σημαίνουν αυτές οι ομάδες και πώς θα λειτουργούν. Καταρχήν δεν θα έχουμε μόνιμες ομάδες δεν θα υπάρχει κάπου στις Βρυξέλλες μια μόνιμη ομάδα που θα ε, περιμένει στο τηλέφωνο. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας σε εθνικούς φορείς και θα κινητοποιούμαστε για συγκεκριμένα καθήκοντα. Σκεφτόμαστε για παράδειγμα κάποιες είτε προγραμματισμένες δραστηριότητες ή κάποιες κατεπίγουσες δραστηριότητες, έκτακτες που θα πετήσουν ταχύ αντίδραση. Άλλη λοιπόν παραστεί ανάγκη, και τα κράτη-μέλη το ζητήσουν, μπορούμε να έχουμε άμεση κινητοποίηση μιας τέτοιας ομάδας. Πάντως, τέτοιου είδου ομάδες ε, κυβερνοασφάλειας είναι εξορισμού λίγο μελίστα. Θα είναι επταμελής, οκταμελής το πολύ. Και μια τέτοια ομάδα, έστω και με 7-8 άτομα, μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Και το λέω γιατί πολλές χώρες, ακόμη και στην αρχική φάση των συζητήσεων, για τη συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες μας επισήμαναν το πρόβλημα των ανθρώπινων πόρων και είπαν ότι δεν έχουμε προσωπικό. Και εγώ, εμείς τους είπαμε, μπορεί να βάζετε έναν στην ομάδα, αλλά ουσιαστικά παίρνετε επτά. Και είναι πραγματικά πολύ αποδοτική μια τέτοια επένδυση, γιατί επταπλασιάζεται η δύναμη. Επίσης, οι ομάδες κυρίως θα βοηθήσουν τις χώρες μέλη που συμμετέχουν σε αυτό το πιλωτικό σχέδιο, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα βοηθούν και άλλες χώρες μέλη, τα θεσμικά όργανα, τις αποστολές κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και χώρες εταίρους. Τώρα, ποιος συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Όταν ξεκινήσαμε την, το σχεδιασμό της ιδέας, σκεφτήκαμε ότι και δύο-τρεις χώρες να λάβουν μέρος, επιτυχημένο θα είναι το σχέδιο δεδομένης ευαισθησίας Τώρα έχουμε ήδη 7 χώρες που συμμετέχουν στο πιλωτικό αυτό σχέδιο και έχουμε πολύ διαφορετικές χώρες. Μικρές, μεγάλες, μεσές, Φιλανδία, κάτω χώρες, ε, Ισπανία, Ρουμανία, Κροατία, ήδη εξέφρασαν επιθυμία συμμετοχής. Έχουμε και παρατηρητές, Γερμανία, Βέλγιο, Στονία, Σλοβενία και Ελλάδα έχουν, παρατηρούν την πρωτοβουλία αυτή. Οπότε θα έχουμε μια αρκετά σημαντική ομάδα για να ελέγξουμε όλες αυτές τις ιδέες και να τις δοκιμάσουμε. Όλες βέβαια οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κάτω ομοφωνία από τα μέλη της ομάδας. Επίσης θέλουμε να αποφύγουμε επικαλύψεις αυτό είναι δεδομένο. Θέλουμε απλώς να ενισχύσουμε τις τρέχουσες πρωτοβουλίες. Και γι' αυτό θα ήταν σημαντικό να διαφυλάξουμε τη σχέση μας και τη συνεργασία με το ΣΕΡΤΙΓΙΟΥ, την ομάδα αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στη, στην πληροφορική, με τον ΕΝΙΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, με το ΣΥΣΕΡ, ομάδα αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας οι υπολογιστές, αλλά και με το το που έχει τις δικές του ομάδες ε, αντιμετώπισης περιστατικό και θα διδαχθούμε και από την εμπειρία του ΝΑΤΟ. Ένα επιπλέον στοιχείο, γιατί το ΠΕΣΚΟ, η ΠΕΣΚΟ δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία ε, που ανέλευθε πρόσφατα στην Ευρώπη, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που επίσης ε, βρίσκεται στα σκαριά και μακροπρόθεσμα θα έχουμε κάποιο σύνδεσμο με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και μακροπρόθεσμα θα χρησιμοποιήσουμε αναπτύξιμες τέτοιες ομάδες ε, ταχείας αντίδρασης ώστε να έχουν τέτοια κινητά αναπτύξιμα εργαλεία και γι' αυτά θα ζητήσουμε ίσως χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το EDF. Αυτή είναι συντομία μια παρουσίαση περιγραφή ακροθυγής της πρωτοβουλίας της Λιθουανίας και περιμένω με χαρά τις απορίες σας. Ο κ. Γκάλερ, μήπως θέλει να ξεκινήσει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση να πω πολιτικά ότι είμαι υπέρ του να στηρίξουμε αυτό το σημείο ως σχέδιο ΠΕΣΚΟ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε παρόμοια προγράμματα που είχαν ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι το όνομα. Αλλά αν χρειαστεί απαραίτητο θα, το, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Εσείς που ασχολείστε. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι θα μπορούμε να αποφεληθούμε και τις εμπειρίες που υπάρχει στον πολιτικό τομέα ώστε να μεταφερθεί αυτή η εμπειρία από τον πολιτικό στον στρατιωτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μοντή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δύο σύντομες ερωτήσεις και θα ήθελα να μου τις αναπτύξετε για αυτή την εθελοντική συνεργασία. Είπατε ότι ίσως να χρειαστεί να υπάρξει και δεσμευτικού τύπου συνεργασία. Θα ήθελα να το εξηγήσετε περισσότερο αυτό, σε ποιους τομείς δηλαδή. Και η επόμενη ερώτηση, επειδή χρησιμοποίησατε το παράδειγμα με τη Λιθουανία, που έχει ένα έδος ε, κεντρικής απάντησης ή κεντρικοποιημένης απάντησης. Έχοντα υπόψη αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως, ε, ήταν ενδιαφέρον να μας το αναπτύξετε αυτό, δηλαδή πώ ε, λειτουργεί αυτό στα πλαίσια της Λιθουανία και ποια είναι η δική σας εμπειρία. Σας ευχαριστώ. Σλόζη. Σας ευχαριστώ. συγγνώμη με λίγο χρόνο. Το ερώτημά μου σχετίζεται με τη συζήτηση που κάναμε σχέση με το προηγούμενο θέμα και όπου αναφέρθηκαν δηλαδή ε, δυνατότητες πιο επιθετικής άμυνας. Ε, σε αυτήν την περιγραφή του project αναφέρεται ότι τέτοιου είδους ομάδες ταχείας απόκρισης θα πρέπει να ε, στοχεύουν στην ε, ταχεία αναγνώριση ακριβώς και στην ε, αντιμετώπιση και στην άμβληση απειλών. Δεν διάβασα κάτι όμως ό,τι αφορά τη δημιουργία περιττέρω ικανότητων. Θέλετε να το κάνετε, υπάρχει τέτοια πρόθεση, έχει αναγνωριστεί μια τέτοια ανάγκη ή μήπως υπάρχει για παράδειγμα μια απαγόρευση ή δεν υπάρχουν τα σχετικά περιθώρια για διεύρυνση των ικανοτήτων. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ένα γενικό ερώτημα σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας αυτού του μηχανισμού. Διαβάσαμε ποια κράτη-μέλη συμμετέχουν εδώ υπό την ηγεσία της Λιθουανίας και διάβασα από εκεί και με το ότι υπάρχουν πέντε κράτη-μέλη παρατηρητές. Ε, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ποια είναι τα δικαιώματα που έχουν αυτοί οι παρατηρητές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι είναι ανταπόκριση σε κυβερνοαπειλέ. Δηλαδή, ποιο ρόλο παίζουν σε αυτό το μηχανισμό οι πέντε παρατηρητέ. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και γίνεται και σημαντικότερο επειδή φαίνεται ότι οι μελλοντικοί πόλεμοι θα είναι κυρίως μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή και οι επίγειες δυνάμεις θα χρειαστούν μόνο για να καταλάβουν στο τέλος την νικημένη χώρα και τα πλέπα θα γίνουν ε, από τον κυβερνοχώρο. Θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Καταρχάς το γεγονό ενδεχομένω αναφέρθηκε προηγουμένω δεν ξέρω βέβαια, αλλά πέρσι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αποφάσισαν να εντάξουν την επίθεση του κυβερνοχώρου ως ε, ρήτρα στο άρθρο 5 για αμοιβαία αρρωγή, το οποίο είναι σημαντικό γιατί η κυβερνοεπίθεση σε μια χώρα σημαίνει ότι είναι επίθεση εναντίον όλου του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι το νέο στο δυτικό κόσμο μεταξύ δυτικών συμμάχων και θα πρέπει να τονίσω το ότι παρόλο που στη συνθήκη της Λισαβόνας είχε θεσπιστεί, αν θυμάστε, το 2009 στο άρθρο 42.7 αυτή η ρήτρα αμοιβαίας ε, αμυντικής αρρωγής Τώρα έχουμε τη θέσπιση και της ε, κυβερνοεπίθεσης η οποία θα πρέπει να θεωρείται ως επίθεση όλων των χωρών μελών και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει μελλοντικά αν θέλουμε να έχουμε μια επιτυχή ΠΕΣΚΟ και μια επιτυχή αμυντική ένωση μέχρι το 2025. Αν το επιθυμούμε αυτό τότε προσεκτικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κυβερνοπόλεμο γιατί είναι αναπόσπαστο τμήμα της προσπάθειάς μας να προστατεύσουμε τις χώρε και τους πολίτε μας στο μέσο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε ζητώντα από τον εισηγητή να απαντήσει στα ερωτήματα και να σχολιάσει αυτά που είπαν τα μέλη της Επιτροπής μας. και οι συνάδελφοι μπορεί να θέλουν και το λόγο αργότερα. Θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω μία προς μία. Αν δεν σας καλύψω, πείτε μου. Καταρχάς, για το στρατιωτικό και το πολιτικό σκέλος και πώς μπορούμε να αποφεληθούμε από την εμπειρία στο πολιτικό σκέλος. Νομίζω ότι εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η πρωτοβουλία, παρόλο που η ΠΕΣΚΟ είναι στρατιωτική πρωτοβουλία και καταρχάς θα έπρεπε να ασχολείται με θέματα άμυνας. Θεωρούμε ότι ο κυβερνοπόλεμος εμπίπτει εδώ σε αυτό το κομμάτι και το εξετάσουμε βέβαια και θα θέλαμε να δούμε οι συμμετέχουσες χώρες μέλη ποιους θα στείλουν δηλαδή αυτές τις πολιτικο στρατιωτικές ε, υπηρεσίες μπορεί να είναι κάποιος στρατιωτικός που μπορεί να οριστεί αλλά θα το αναπτύξουμε αυτό ξαναλέω και στο εσωτερικό των ομάδων αυτών θα υπάρχει ένα συμπειρογνώμα για αυτά τα πολιτικο-στρατιωτικά θέματα για την κυβερνοασφάλεια και το αντίστοιχο πολιτικό κομμάτι. Ναι, βέβαια, το εξετάζουμε σε συνεργασία με το δίκτυο σες e, το οποίο αποτελεί μια πιλωτική πρωτοβουλία χωρών για αυτά τα θέματα. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι όλοι προσβλέπουμε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν γρήγορα και επιθετικά. Αλλά στην Ένωση ξεκινάμε με την ανταλλαγή πληροφοριών, με την δυνατότητα ε, επικοδομής ανθεκτικότητας και προσπαθούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Και αν υπάρξουν αντίστοιχε αποφάσεις μελλοντικά, ευχαρίστω θα τις στηρίξουμε. Μετά υπάρχει και το θέμα των εθελοντικών και δεσμευτικών δεσμεύσεων, λέει ο μιλητής. Όλα αυτά που κάνουμε στην ΠΕΣΚΟ είναι εθελοντικά και θέλουμε να κάνουμε βέβαια περισσότερα. Όμως, από ό,τι ξέρετε, η ίδια η ΠΕΣΚΟ είναι κάτι περισσότερο από τις αμοιβέ δεσμεύσεις. Δηλαδή, χωρίς την ΠΕΣΚΟ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά η ΠΕΣΚΟ θα μπορούσε να παράξει, να προκαλέσει περισσότερα από αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η απάντηση λοιπόν είναι ενδεχομένως ότι όντως η ανάπτυξη αυτής της ευθύνης είναι σε θελοντική βάση. Όμως, από τη στιγμή που αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, αυτό γίνεται κάτι πιο δεσμευτικό στα επίπεδα συνεργασίας. Και νομίζω αυτό είναι το σκεπτικό, αυτή είναι η λογική των παροτρήσεων μας προς τις χώρες μέλη για, ένα πιο, για τη μετάβαση από ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον σε μια πιο δεσμευτική συνεργασία. Μετά για τις εθνικές μας εμπειρίες από το Γενάρη μόνο έχουμε αντίστοιχε εμπειρίες οπότε δεν έχουμε πολλά να μεταδώσουμε και η απόφαση γιατί για ποιο λόγο δηλαδή αποφασίσαμε να κάνουμε αυτά που κάναμε, είναι επειδή καταλάβαμε ότι μας λείπουν οι κυβερνοπόροι για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων. Έχουμε μικρότερες υπηρεσίες. Έχουμε αυτή ας πούμε, που ασχολείται ας πούμε, με θέματα κυβερνητικά, άλλοι που ασχολείται με θέματα στρατιωτικά ή πολιτικά και αν κάνουμε κατακαιρματισμό των πόρων και υποδομής. Έχουμε αυτό που έχουμε στη δικιά μας την περίπτωση θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τις δαπάνες ώστε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους πόρους. Πάντως ελπίζουμε ότι σε περίπου ένα χρόνο θα έχουμε εμπειρία να μοιραστούμε με τις χώρες μέλη για αυτά τα πράγματα. Μετά για την επιθετική μας ικανότητα. Νομίζω ότι εξαρτάται από τις χώρες μέλη το πώς θα αναπτυχθεί αυτή η πρωτοβουλία. Είναι σαφές ποιο είναι το σημείο κίνησης, να υπάρχει δηλαδή καλύτερη απάντηση η ανάλυση και η μετρίαση των απειλών στον κυβερνοχώρο, αλλά αυτό ξαναλέω εξαρτάται από τις ε, χώρες μέλη και αυτό συμβαδίζει με το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Ακόμα και να ξεκινήσουμε συζητήσει για την κυβερνοασφάλεια, πρέπει να υπάρχει βέβαια εμπιστοσύνη. Το να ξεκινήσουμε συζητήσει για θέματα επιθετικά, πάλι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Το συζητάμε ε, αυτά, ε, αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια, αλλά αυτά είναι πρωτοβουλίες άμυνας και καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει και το στοιχείο της μυστικότητας επειδή οι χωρισμένοι αναπτύσσουν τη δικιά τους ικανότητα απάντησης. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για το μέλλον. Μετά, για τους παρατηρητές στις ομάδες μας. Γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τους παρατηρητές της ΠΕΣΚΟ. Οπότε δεν αφορά μόνο το δικό μας πρόγραμμα αυτό. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει καθεστώς παρατηρητή και το κατά πόσο συμβάλλουν στις πρωτοβουλίες. Υπάρχει πάντως συνένεση για το να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο καθεστώς και οι χώρες μέλη με αυτόν τον τρόπο ζητούν περισσότερες πληροφορίες και ευκολύνουν τη διαδικασία ώστε τελικά να γίνουν χώρες μέλη που συμμετέχουν δηλαδή σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς βεβαίως καλωσορίζουμε, είναι ευπρόζεκτοι οι παρατηρητές από μια ομάδα χωρών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ως μέλη στα προγραμματά μας. Έχουμε διάλογο με αυτές τις χώρες, όταν όμως ε, είμαστε στην λειτουργική φάση των προγραμμάτων ή στη χάραξη των προγραμμάτων, αυτό αφορά αποκλειστικά τις χώρες που συμμετέχουν στα προγράμματα. Και τέλος, σημείωσα άλλη μια ερώτηση για το ΝΑΤΟ και το άρθρο 5 σε σχέση με τον κυβερνοπόλεμο και τη ρήτρα αμοιβαίας αρρωγής. Εγώ με αυτή την άποψή σας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υποβάλαμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί εδώ ακριβώς έχουμε κάνει την προστασία της Ευρώπης που σημαίνει προστασία των πολιτών της. Εμείς δεν το προσεγγίζουμε ως κάτι που αποτελεί μια επικάλυψη σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Εμείς θεωρούμε ότι αντίθετα το ενισχύει και κάτι σημαντικό που διαχωρίζει τις συζητήσεις στο ΝΑΤΟ από τις συζητήσεις στην Ένωση είναι ότι το ΝΑΤΟ εμπλέκει περισσότερο παράγοντες ε, στρατιωτικούς και ανταπόκριση στο, στις καιρούν Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα της διασύνδεσης στρατιωτικού με το, πολιτικού, με το πολιτικό σκέλος. Και σε μια κατάσταση κρίσης ο στρατιωτικός παράγοντας θα πρέπει να είναι σε θέση και ικανός να ανταποκριθεί σε αυτές τις κυβερνό Αλλά σε καιρό ειρήνης, παρόλο που έχουμε κυβερνοεπιθέσεις ε, σε καθημερινή βάση και σε μεγάλους αριθμούς, αυτοί οι στρατιωτικοί παράγοντες θα πρέπει να συνεργάζονται με τους πολιτικούς παράγοντες και να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για καταστάσεις καθημερινές και πρακτικές. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε κι εμείς όταν αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα συνεργασίας, δηλαδή μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού παράγοντα, ώστε να έχουμε την κατάλληλη απάντηση. Σας ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλος κανεί το λόγο, οπότε να υποβάλω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Το θέμα του κυβερνοχώρου εντοπίστηκε ως τομέα συνεργασίας Ευρωπαϊκή Ένωσης ΝΑΤΟ. Και εμείς συνεχώς επισημαίνουμε την ανάγκη αποφυγή των επικαλύψεων και στον στρατιωτικό τομέα. Έχετε σκεφτεί πώς στα πλαίσια της δικής σας πρωτοβουλίας θα συνεργαστείτε με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι αμοιβαίας δέσμευσης και συνεργασίας ώστε να γίνει ένας επιμερισμός του έργου και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Δεύτερον, Έχετε σκεφτεί τι είδους δράσεις θα συμπεριλάβετε στο σχέδιό σας. Ανάλογα με τους δράστες των επιθέσεων. Γιατί είναι διαφορετικό κάθε φορά το προφίλ του δράστη. Και ανάλογα με τις διαφορές αυτές ε, θα επεξεργαστείτε διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης ανάλογα με το αν πρόκειται για κρατικό φορέα ή όχι γιατί και εκεί θα πρέπει να ξεπεράσετε κάποιες δυσκολίες. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ξέρετε όντως που ε, βρίσκονται δυσκολίες ό,τι φορά τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Αυτό επηρεάζει και τη δική μας συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Πάντως, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και να διδαχθούμε από την εμπειρία του ΝΑΤΟ. Αλλά σε αυτό το στάδιο πιο επίσημη συνεργασία δεν είναι εφικτή. Παρόλο που, όπως είπατε, ο κυβερνοχώρος έχει εντοπιστεί ως πιθανός τομέα συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, αλλά περισσότερο αφορά την ευαισθητοποίηση της κατάστασης και τη κοινή αντίληψη των απειλών περισσότερο. Πάντως πιστεύω ότι και οι δικές μας ομάδες θα ε, εποφεληθούν από μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ή την αντίστοιχη ομάδα του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας σε υπολογιστές. Πάντως, επί του παρόντος δεν βλέπουμε υπάρχει δυνατότητα για επίσημους τυπικούς δεσμούς με το ΝΑΤΟ. Πάντως σίγουρα θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο την εμπειρία του ΝΑΤΟ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των ε, δραστηριοτήτων μας ανάλογα με τους ε, δράστες των κυβερνοεπιθέσεων. Καταρχήν, ε, η πρώτη αντιμετώπιση γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και σε περίπτωση κρίσης, ε, είναι δύσκολο μόνο το ένα κράτο μέρος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και σε τέτοια περίπτωση μιλούμε για κινητοποίηση της ομάδας. Αλλά μιλούμε για μεγαλύτερη κρίση, για ευρύτερη. Αλλιώ, όταν είναι μικρή εμβέλεια, ένα κράτο μέρο μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει. Αλλά όταν μιλάμε για τέτοια κρίση, πολύ σπάνια κρατικό φορέα είναι ο δράστης ε, μάλλον, ε, για μεγάλη κρίση, μάλλον κρατικός φορέ βρίσκεται πίσω από τους δράσεις επιθέσεις, γιατί μεμονωμένοι hacker δεν έχουν τέτοιε δυνατότητες. Μερικές φορές κρατικοί παράγοντες ε, δοκιμάζουν ε, και ελέγχουν τα δίκτυά μας. Ο κύριος Φροντσούλικα λυπάμαι που επανέρχομαι με ερώτηση, αλλά πραγματικά δικές ερωτήσεις δίνουν ενάψματα για περαιτέρω συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων. Αν θέλουμε να δώσουμε σάρκα και οστά στην πρωτοβουλία αυτή, και μιλώ για το ΠΕΣΚΟ, Γνωρίζετε το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλά για τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Το άρθρο λοιπόν αυτό προβλέπει ότι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να βοηθήσουν ε, ε, μία άλλη χώρα μέλος που έγινε θύμα ένοπλης επίθεσης στην επικράτειά του. Ένοπλης επίθεσης. Αυτό στο μέλλον θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του συγκεκριμένου άρθρου της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα ήταν αδύνατο να επικαλεστεί κανεί κυβερνοεπίθεση για να ζητήσει συνδρομή όταν έχουμε ένα τέτοιο άρθρο που μιλά μόνο για ένοπλη επίθεση. Δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημη διαδικασία για το αίτημα αρρωγή. Βέβαια υπάρχει το ιστορικό, γιατί η Γαλλία επικαλέστηκε το άρθρο αυτό το 2015 μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι ξεκινώντας διμερείς συζητήσεις στα κράτη-μέλη, χωρίς όμως ε, ένα σαφές ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο συνεργασίας. Εκεί κάθε χώρα είχε διαφορετική γνώμη και προσέφερε με διαφορετικό τρόπο ε, συνεργασία ή βοήθεια εμπειρογνώμονες, ε, η αποστολή περισσότερων στρατευμάτων στη Συρία ή το Ιράκ βοηθώντας τα γαλλικά στρατεύματα στην Αφρική, στο Μαλί για παράδειγμα ή αλλού, ώστε να μπορέσουν οι Γάλλοι να στείλουν στρατεύματα τους σε άλλες χώρες. Αλλά αυτά όλα αυτά πρέπει να τα προσδιορίσουμε με σαφήνεια, θέλουμε μια πραγματικά μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, μια πραγματική πέσκο. Δεν μπορούμε να επαφιόμαστε μόνο στις διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών μελών. Αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν προαιωνίζεται ε, λαμπρό μέλλον για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας. Έχετε το λόγο. Θέλετε να σχολιάσετε. Συμφωνώ, συμφωνώ ότι είναι κάπως παρακινδυνευμένο αυτό. Και όντως εμείς επιδιώκουμε αμοιβαία αρρωγή και το λέμε στον τίτλο του σχεδίου γιατί μακροπρόθεσμα προσβλέπουμε σε αμοιβαία αρρωγή πραγματικά μεταξύ των συμμετεχών των κρατών μελών. Και για μας και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να προστατεύει την Ευρώπη και να παρέχει αμοιβαία αρρωγή μεταξύ των κρατών. Βέβαια είναι διαφορετικές ερμηνείες που έχουν δοθεί στο άρθρο αυτό, ιδιαίτερα μετά την επίκληση του από τη Γαλλία. Σίγουρα η υποχρέωση αρρωγής αφορά τα κράτη-μέλη, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, πολύ καλή αυτή η ιδέα για την Επιτροπή μας, κυρία Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε εμείς κάλλιστα να κατατήσουμε έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Αμοιβαίας Άμυνας. Έτσι θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε με τη δική μας έκθεση στην ε, σκέψη και τη συζήτηση που γίνεται. Πολύ καλή ιδέα, αλλά θα την αφήσουμε για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Γιατί έχουμε καθορίσει το νομοθετικό μας έργο μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας ε, και εμείς δεν μπορούμε να προσθέσουμε νέα θέματα. Πάντως συμφωνώ ότι είναι μείζον ζήτημα και στο μέλλον θα πρέπει να εξεταστεί. Μάλιστα, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να χειροκροτήσουμε τον καλεσμένο μας. Και παραμένετε στην αίθουσα γιατί έχουμε και άλλο σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη που θα γίνει όμως ε, και κλεισμένο των θυρών. Πρόκειται για την επίθεση που έγινε στο Σάλσμπερι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη χρήση ενός νευροτοξικού, νευροπαραλυτικού αερίου στο Σόλσμπερι. Καλεσμένος μας είναι ο Βρετανός πρέσβης στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Πολ Τζόνστον. Παρακαλώ, μόνο οι ευρωβουλευτέ δικαιούνται να παραμείνουν στην αίθουσα, μια και πρόκειται για και κλεισμένων των θύρων συνεδρίαση. Οι σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων και βοηθοί δεν επιτρέπεται να παραμείνουν. Εκπρόσωποι επίση των θεσμικών οργάνων μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα. Παρακαλώ η Γραμματεία να φροντίσει να παραμείνουν μόνο οι δικαιούνται να είναι παρόντες.